Uh, Εξοχοτάτη, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά αρχίζουμε τη συνεδρίαση και σας καλωσορίζουμε κυρία Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε δε που βρήκατε το χρόνο να μας επισκεφθείτε. Κυρία Υπουργέ, Λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης η χώρα σας, το Πακιστάν, βρίσκεται στο προσκήνιο της καταπολέμησης των ακρεωτήτων, όχι μόνο στα σύνορά της αλλά και εσωτερικά. Η κυβέρνησή σας προσπαθεί να εφαρμόσει την εφταξία και να καθησυχάσει τις εντάσεις εσωτερικές και εξωτερικές. Ομαλοποιήσατε τις σχέσεις σας με την Ινδία και αυτό επιτέχθηκε γιατί και οι δύο πλευρές αποφάσισαν οι σχέσεις τους να μην κυριαρχούνται μόνο από τη διαμάχη για το Κασμίρ, την Πενταποταμία. Και γνωρίζουμε επίσης ότι και οι σχέσεις σας με τα δεν είναι πολύ εύκολες και ότι η περίπτωση να φύγουν από το Αφγανιστάν οι ξένες δυνάμεις θα μπορούσε να θέσει ορισμένα ερωτηματικά και ανησυχίες. Κυρία Υπουργέ, η κυβέρνησή σας πρέπει να πετύχει το δύσκολο καθήκον να καταπολεμήσει την τρομοκρατία και τις ακρότητες, αλλά και να καθησυχάσει τους φόβους του λαού. Ως η πρώτη γυναίκα Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν γνωρίζετε ότι είναι σύγχρονη χώρα το Πακιστάν χώρα στην οποία οι γυναίκες σιγά σιγά απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρας. Με μεγάλη χαρά λοιπόν σας δίνω το λόγο για την παρουσίασή σας και μετά φαντάζομαι ότι θα ακουστούν και ερωτήσεις. Σας κατευχαριστούμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να πω ευθύς εξ αρχής πως ε, αυτό η σημερινή συνάντηση για εμένα και τη χώρα μου είναι μια μεγάλη ευκαιρία ευκαιρία να έρθουμε εδώ πέρα και να αναφέρουμε τις προκλήσεις που έχουμε στο Πακιστάν και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και στο Πακιστάν και σε ολόκληρη την περιοχή με κάπως περισσότερες λεπτομέρειες. Πρώτα απ' όλα, κυρία Πρόεδρε, νομίζω πως αναφερθήκατε σε κάτι το σημαντικό και χαίρομαι που το αναγνωρίζετε στα τέσσερα τελευταία χρόνια όπου έχουμε δημοκρατική διακυβέρνηση στο Πακιστάν είχαμε μία σαφή έμφαση που χαίρομαι πως ε, σημειώνεται η αναγνώριση δηλαδή του ότι η ειρήνη ε, στο εσωτερικό θα πρέπει να ξεκινήσει από την ειρήνη στο εξωτερικό. Οπότε αν δείτε την εξωτερική πολιτική του Πακιστάν είχαμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση το ότι με μεγάλο ζήλο ερχόμαστε σε επαφή με τους γειτονές μας. Πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να ειρηνεύσουν τα σύνορά μας, είτε είναι με την Ινδία η οποία τυχαίνει να είναι μια χώρα με την οποία έχουμε βεβαίως 60 χρόνια έχθρας, πολέμων, τριών πολέμων, συγκρούσεων, αλλά οι λόγοι βεβαίως είναι γνωστοί. Έχουμε δαφικές διαφορές μεταξύ των οποίων το Κασμίρ, Τζαμού και Κασμίρ, αλλά αποφασίσαμε πως είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στην Ινδία όπου δεν θα κάνουμε πόλεμο, αλλά θα προσπαθούμε το κάθε ζήτημα να το λύνουμε στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Και έτσι αποφασίσαμε να αναστρέψουμε μια πολιτική 40 ετών ε, με την οποία δεν είχαμε εμπορικές σχέσεις με την Ινδία και βεβαίως είχαμε έναν θετικό κατάλογο αντικειμένων ε, στα οποία μπορούσαμε να εμπορευτούμε. Το αντιστρέψαμε αυτό και τώρα έχουμε πλήρως ομαλές εμπορικές σχέσεις και ελπίζουμε έτσι πλέον να έχουμε αμοιβαία συμφέροντα έτσι ώστε οι άνθρωποι στην Ινδία και στο Πακιστάν να επιφελούνται από το κοινό μας μέλλον. Ταυτόχρονα, αν κοιτάξετε προς μας... Το Αφγανιστάν είναι μια χώρα με την οποία είχαμε πολύ ε, διαφορετικές σχέσεις από ό,τι με την Ινδία. Το Αφγανιστάν είναι μια χώρα όπου παραδείγματο χάρη τα, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ε, έχουμε υποδεχτεί τρία εκατομμύρια Αφγανούς πρόσφυγες στο εδαφός μας. Ήμασταν φιλόξενοι, ανοίξαμε τα σχολεία μας, ε, τις πόλεις μας και εδώ και τρεις δεκαετίες και οπωσδήποτε την τελευταία δεκαετία η αστάθεια του Αφγανιστάν ε, περνάει τα σύνορα και διαχέεται και στη χώρα μας συνεχώς. Ένα άλλο μάθημα το οποίο διδασκόμαστε είναι πως, από την ιστορία, είναι πως δεν μπορεί να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα στο Πακιστάν αν δεν υπάρχει ειρήνη και σταθερότητα στο Αφγανιστάν. Έχουμε σύνορα μήκους 2.600 χιλιόμετρων, τα οποία διασχίζουν κάθε μέρα 50.000 άνθρωποι, 56.000 άνθρωποι κάθε μέρα. Οπότε ό,τι συμβαίνει στο Αφγανιστάν μας επηρεάζει άμεσα. Η πολιτική που έχουμε με το Αφγανιστάν είναι πως ο μόνος κανόνας ε, ε, που έχουμε είναι πως ο ρόλος μας είναι να ε, διευκολύνουμε την ειρήνη, την σταθερότητα και την ασφάλεια. Δεν σκοπεύουμε να πάμε παραπέρα. Και στο πλαίσιο αυτό έχουμε κάνει μεγάλα ανοίγματα στο Αφγανιστάν. Ο πρόεδρος μας όταν ορκίστηκε κάλεσε μόνο τον κύριο Καρζάη να παραστεί στην ορκομοσία του ως ξένο αξιωματούχο και ήταν ακριβώς το μήνυμα πως θέλουμε να έχουμε σχέσεις μαζί τους ως ε, ισότιμες χώρες. Ε, και πάλι σας λέω, έχω πάει στο Αφγανιστάν περισσότερο οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο και υποδέχτηκα την Παρασκευή των υπουργών Εξωτερικών τους και βεβαίω θα ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος Καρζάη στη Νέα Υόρκη, δηλαδή συζητήσεις για την ε, συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας. Δηλαδή, καθώς υπάρχει μια μετάβαση στο Αφγανιστάν και οι ανησυχίες για ένα κενό ασφαλείας που υπήρχαν είτε από μας είτε από αλλού, οι θεσμικές, διπλωματικές, πολιτικές έπαφες μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν θα είναι εξαιρετικά σημαντικές. Οπότε θα δημιουργηθούν αυτές οι θεσμικές επαφές στο μέλλον. Οπότε, ναι, αν θέλετε να δείτε πού πηγαίνει το Δημοκρατικό Πακιστάν, νομίζω πως η εξωτερική πολιτική είναι ένας καλός τρόπος. Αλλά ας πάμε πέρα από την εξωτερική πολιτική, γιατί μίλησα βεβαίως για ε, ισχυρές με ολόκληρη την περιοχή. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο σε εσά μοιάζει χαοτικό, γιατί οι ειδήσει που έρχονται από το Πακιστάν μοιάζουν χαοτικές, είναι θεσμικά όργανα του Πακιστάν που βρίσκουν τον συνταγματικό τους ρόλο. Είτε είναι το Κοινοβούλιο, είτε είναι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, είτε είναι η κοινωνία των πολιτών, είτε είναι τα ΜΜΕ, είτε άλλα θεσμικά όργανα. Όλοι τώρα βρίσκουν μια θεσμική ισορροπία που δημιουργήθηκε με το Σύνταγμα 1973. Θέλω τώρα να επισημάνω κάποια επιτεύγματα της δημοκρατικής κυβέρνησης των τελευταίων ετών. Το σημαντικότερο νομίζω είναι πως όταν αναλάβαμε καθήκοντα ο πρόεδρος Σαρντάρη είπε πως ο πόλεμος αυτός ο οποίος στο, εμείς θεωρούμε ότι μας επιβλήθηκε από την Δύση δεν μπορεί να είναι πόλεμος κάποιου άλλου όταν σκοτώνονται τα δικά μας παιδιά και το δικό μας πληθυσμό και τους δικούς μας στρατιώτες. Οπότε αυτό το οποίο κάνουμε, δηλαδή να κάνουμε δικό μας τον αγώνα κατά των ε, ακραίων στοιχείων ήταν κάτι το άνευ ε, προηγουμένου και έτσι μέσω του Κοινοβουλίου μπορέσαμε να κάνουμε σημαντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Βαζιριστάν και στο Μολεγάν. Γιατί όταν ανέλαβε καθήκοντα η κυβέρνησή μας ε, γύρω στο 30% των ε, φιλετικών περιοχών ήταν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης. Σήμερα είναι γύρω στο 70%. Βλέπουμε λοιπόν τι μπορεί να επιτύχει η δημοκρατία εάν ξέρει το τι είναι καλύτερο για τον ε, λαό και μας επιτρέπει να κάνουμε το σωστό για το κράτος και για το λαό. Κατόπιν, ε, υπήρχαν πάρα πολλά λάθη που έπρεπε να διορθωθούν στο Πακιστάν, γιατί το Πακιστάν ε, είχε συσταθεί ως ομοσπονδία με περιφέρειες οι οποίες θα είχαν δικούς τους πόρους ε, και θα μπορούσαν έτσι να έχουν κάποια αυτοδιοίκηση και να αναπτυχθούν και να αναπτύξουν τη χώρα τώρα. Με επί σειρά ετών και κυβερνήσεων ε, είχε αλλάξει το Σύνταγμα Πολάκης από τις πολλές στρατιωτικές κυβερνήσεις. Τώρα, όταν αναλάβαμε εξουσία στο Κοινοβούλιο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε βέβαια, αν δεν έχει κανείς πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, ε, ξέρετε, μια συμμαχική κυβέρνηση είναι λιγότερο αποτελεσματική. Και ακόμη περισσότερο αν δεν έχει κανείς ε, ισχυρή πλειοψηφία ούτε ως ε, συνασπισμός. Καταφέραμε όμως να κάνουμε τρεις αλλαγές στο Σύνταγμα που απαιτούσαν ε, πλειοψηφία δύο τρίτων. Η πρώτη επανέφερε το Σύνταγμα του 1973 και έδωσε στις ε, περιφερειές τα δικαιώματά τους. Η δεύτερη και τρίτη αλλαγή του Συντάγματος ενίσχυσε περαιτέρω την εκλογική επιτροπή του Πακιστάν και τους τρόπους για να γίνει αυτό. Οπότε αυτό το οποίο συνέβη είναι πως τα ρήγματα που υπήρχαν εντός του Πακιστάν μεταξύ των περιοχών εντός των περιοχών και μεταξύ περιοχών και ομοσπονδίας ξεκαθάρισαν και έτσι η ευθύνη και οι πόροι πήγαιναν τώρα στην ίδια αρχή. Δηλαδή αν η εκπαίδευση και η υγεία ήταν αρμοδιότητα των περιφερειών είχαν και τους πόρους. Σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Επίσης η Εθνική Χρηματοδοτική Επιτροπή είναι το μέσο μέσα στον οποίο γίνεται η διανομή των πόρων. Αλλά δεν είχε συσταθεί για 20 ε, χρόνια ούτε με κοινοβουλευτική ούτε με στρατιωτική κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε πως είχε φτάσει η ώρα να συσταθεί, να δώσει περισσότερα λεφτά στις περιφέρειες και άρα έτσι υπήρχε αυτός ο μηχανισμός αναδιανομής των πόρων. Επίσης κάτι το οποίο είναι σημαντικό και ξέρω πως σας ανησυχεί και εμείς χαιρόμαστε για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική προστασία ότι είναι κάτι το σημαντικό γιατί εμείς θεωρούμε πως είστε παραδείγματα κοινωνιών για το Πακιστάν. Κοινωνίες που προστατεύουν τους αδυναμούς. Δυστυχώς στη χώρα μου και σε χώρες σαν μου χρειάζεται νομοθεσία για να προστατευτούν οι αδύναμοι και μετά βέβαια η κοινωνία να τα οικοδομήσει αυτά. Εγώ είμαι υπερήφανη που εκπροσωπώ μια κυβέρνηση που ανέλαβε την ευθύνη να προστατεύσει τους αδύναμους του Πακιστάν. Θα θέλαμε να είμαστε μια χώρα κοινωνικής πρόνοιας, όμως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τους πόρους Τι κάναμε λοιπόν. Παρά τους πενιχρούς πόρους που έχουμε, είπαμε πως το κράτος πρέπει να προστατεύει τους πιο ευπαθείς. Τι κάναμε λοιπόν. Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα στήριξης εισοδήματος Μπενιζήρ, το οποίο δίνει οικονομική στήριξη και ασφάλιση υγείας ε, στους πιο αδύναμους και δυνατότητες απασχόλησης κτλ. Και για να κερδίσουμε περισσότερο από αυτό, τι κάναμε. Αντί το ποσό αυτό να πάει στον άντρα της οικογένειας, πήγαινε στη γυναίκα της οικογένειας. Και έτσι αυξήθηκε το κύρος της γυναίκας στο σπίτι της, γιατί πλέον ήταν μια πηγή εισοδήματος. Επίσης, είμαστε υπερήφανοι γιατί κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια μπορέσαμε να κάνουμε πολύ μεγάλα βήματα για την προστασία των γυναικών. Περάσαμε τρία, τέσσερα νομοσχέδια και μας ενδιαφέρει η προστασία των γυναικών κατά της οικογενειακής βίας στην εργασία και για πρώτη φορά έχει συσταθεί μια ανεξάρτητη ομάδα, επιτροπή μάλλον ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία ασχολείται με συναφή ζητήματα. Πρόκειται για ε, σοβαρά βήματα τα οποία επιτελέσαμε και θα ήθελα να απαντήσω και ενδεχόμενες ερωτήσεις δικές σας, αλλά θεωρώ ότι το Πακιστάν αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις έχει να αντιμετωπίσει και πολύ περισσότερες και προσπαθήσαμε ενεργά να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ, για αυτή την εισήγηση, η οποία είναι άκρος διαφωτιστική. Τώρα θα δώσω, θα δώσω το λόγο στον κύριο Σαλαφράνκα, τον συντονιστή από την ομάδα του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω την Υπουργό. Περιμένω να βάλει τα ακουστικά της. Ευτυχώς έχουμε χρόνο σήμερα. Για να eh, Θα ήθελα εξ ονόματος του ΕΛΚ να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω διότι βρίσκεστε εδώ να μας εκθέσετε τις απόψεις σας. If you could mute please. It's working. Sí, eh, Σας ε, ευχαριστούμε, Υπουργέ, για την ε, παρουσία σας εδώ εξ ονόματος ε, της ομάδας μου. Οι Βρυξέλλες δυστυχώς έχουν πληγεί από κακοκαιρία, γι' αυτό και δεν είμαστε πολυπληθής εδώ ομάδα και επιτροπή, αλλά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας. Θα ήθελα να αναφερθώ στο, στο πολιτικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα σας. Μιλήσατε εσείς για τις κινήσεις των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ εκτελεστικού και νομοθετικού και θα θέλαμε να μας μιλήσετε για την πολιτική κατάσταση εν ώψη των επόμενων εκλογών την επόμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος. Κυρία Υπουργέ, ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο ενέκρινε ένα ψήφισμα για τη νέα Μαλάλα η οποία είχε απειληθεί με θάνατο από τους ε, Ταλιμπάν. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς ε, μπορείτε να ε, εξασφαλίσετε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, πώς αντιμετωπίζετε τις απειλές. Μας ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα της γυναίκας και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και γενικότερα, ποια είναι τα μέτρα που θα λάβει υπόψη, που θα λάβει μάλλον η κυβέρνησή σας. Είπατε ότι όταν η κατάσταση αποσταθεροποιείται στο Αφγανιστάν έχει άμεσες συνέπειες. Μιλείς, στη χώρα σας μιλήσατε για τα κοινά σύνορα των, ε, που, είναι δυο, που ενέρχονται σε 2.500 χιλιόμετρα και θα ήθελα να ρωτήσω πώς ε, αντιμετωπίζετε την κατάσταση μετά την απόσυρση των ε, διεθνών δυνάμεων που θα επισυμβεί το 2014. Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί, θα υπάρξει μία επιπρόσθετη αστάθεια ή όχι. Επίσης, πώς θα αντιμετωπίσετε τη μεγάλη πρόκληση της απειλής των Ταλιμπάν και πώς μπορείτε να συνδράμετε έτσι ώστε να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε έμπρακτα αυτή την απειλή. Θέλετε να απαντήσετε άμεσα ή να... Ε, ή θέλετε να γύρω ερωτήσουν. Όχι, να απαντήσετε. Εντάξει, έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Ωραία. Πρώτα απ' όλα αναγνωρίζω, θα έπρεπε να το είχα κάνει από την αρχή, ποια είναι η βοήθεια που μας χορηγεί η Ένωση. Είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έρθει σε βοήθεια προς το Πακιστάν σε πολλά θέματα με την ενεργοποίηση των ρητρών ATP στις συμφωνίες. Είναι σοβαρός τρόπος βοήθειας μιας χώρας που απειλείται από την τρομοκρατία και που την καταπολεμεί από την πρώτη γραμμή. Τώρα, μιλήσατε γενικά για το πολιτικό κλίμα στο Πακιστάν. Τα τελευταία 60 χρόνια της ύπαρξής του, το Πακιστάν ζούσε δημοκρατικά. Αυτό δείχνει ποιο είναι γενικά το πολιτικό κλίμα. Πάντοτε βέβαια υπάρχουν ομάδες και κόμματα που έχουν διαφορετικούς στόχους μεταξύ τους, αλλά πολλά από αυτά τα κόμματα που αντιμάχονται το ένα το άλλο στις εκλογές συνεργάστηκαν όχι μία φορά αλλά τρεις για να εγκριθούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούν πλειοψηφία δύο τρίτων και αυτό δείχνει την πολιτική οριμότητα που υπάρχει στο πακιστανικό πολιτικό σύστημα όταν χρειάστηκε να γίνει μια στρατιωτική επιχείρηση, αυτό έγινε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των πολιτικών κομμάτων. Άρα μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί η πολιτική ζωή όρημα. Επίσης μιλήσατε για τη διαφορά νομοθετικού και εκτελεστικού. Φαντάζομαι εννοείται από τη μία το κοινοβούλιο και από την άλλη την κυβέρνηση. Οι σχέσεις είναι πολύ καλές. Πολλά από τα σημαντικά νομοσχέδια που χρειάστηκαν πέρασαν φυσικά με την έγκριση του Κοινοβουλίου. Μετά μιλήσατε για την Δεσποινίδα Μαλάλα και την προστασία που πρέπει να της χορηγηθεί. Θα της χορηγηθεί αυτή τη στιγμή είναι σε νοσοκομείο στη ΣΥΠΑ και η κυβέρνηση πληρώνει όλα τα έξοδα. Ακόμη και όταν οι τρομοκράτες την είχαν απειλήσει προηγουμένως, από τότε η κυβέρνηση της πρόσφερε προστασία και ασφάλεια. Σε τρεις τουλάχιστον χωριστές περιπτώσεις. Αλλά αρνήθηκε η οικογένειά της. Φυσικά είναι ευθύνη μας και την παίρνουμε πολύ σοβαρά. Επίσης θέλω να αναγνωρίσετε ότι Όλο το Πακιστάν υποστήριξε την περίπτωση της Μαλάλας και αυτό που ζητούσε και η ίδια να έχει κάθε παιδί το δικαίωμα σε εκπαίδευση και το όραμα του Πακιστάν που αντιπροσωπεύει εκείνη το δέχονται όλος ο πληθυσμός, μόνο μία ελάχιστη μειονότητα διαφωνεί. Είδατε όμως και τι έγινε με την επίθεση. Όλο το Πακιστάν δέχτηκε τις δικές της, το δικό της όραμα για το Πακιστάν. Μετά μιλήσατε για το Αφγανιστάν και πώς βλέπουμε τα πράγματα εκεί. Αν θα υπάρξει δηλαδή περισσότερη σταθερότητα εκεί ή λιγότερη. Δεν μπορώ να σας απαντήσω από τώρα γιατί αυτό εξαρτάται από το τι θα γίνει και πώς θα γίνει μέχρι το 14. Είναι πολύ σημαντικοί οι επόμενοι μήνες. Από τώρα μέχρι το 14 θα δούμε αν μπορεί να μπορέσουν να δημιουργηθούν οι συνθήκες στο Αφγανιστάν ώστε να μην είναι αναστρέψιμος ο εκδημοκρατισμός της χώρας και όλες οι οργανώσεις που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν βία να γίνουν πολιτικές οργανώσεις με ειρηνική και δημοκρατική διαβίωση. Αυτό θα καθορίσει το μέλλον του Αφγανιστάν. Αλλά με καθησύχασε το γεγονός ότι τελευταία άκουσα το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να μου λέει να είστε βέβαιοι ότι δεν θα αφήσουμε φεύγοντας κενό ασφαλεία στο Αφγανιστάν. Αυτό ζητούσαμε και εμείς ως γείτονες. Ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ. Τώρα ο συντονιστής των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών σας καλωσορίζω και εγώ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντοτε χαιρόμαστε όταν βλέπουμε γυναίκες σε υψηλά αξιώματα. Είναι κάτι που μπορεί και για μας να αποτελέσει μάθημα γιατί στο, Υπουργείο, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών θα δείτε ότι είναι όλο άντρες. Συγχαρητήρια λοιπόν. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω ε, ε, ε, θα ήθελα να ρωτήσω πώς επηρεάζει η οικονομική κρίση το Αφγανιστάν, ποιες είναι οι κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζετε. Διότι τα κοινωνικά προβλήματα έχουν άμεση προεπίπτωση στη δυνατότητα των εξτρεμιστών να προσελκύσουν κόσμο. Είπατε ότι σημειώθηκε πρόοδος στην καταπολέμηση του εξτρεμισμού και ότι ο αγώνας αυτός δεν επιβλήθηκε από τα έξω αλλά το ίδιο το Πακιστάν τον ασκεί. Φυσικά δεν γίνεται μόνο με μέτρα ασφαλείας και στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά τι άλλο κάνετε, πώς μπορείτε να επιτύχετε αυτή την αλλαγή και πώς σχετίζεται αυτό και με την παιδεία, διότι όσο πιο μορφωμένοι είναι οι άνθρωποι, τόσο λιγότερο θα ενδιαφέρονται για εξτρεμιστικές στάσεις και δραστηριότητες. Τι μέτρα λοιπόν χρειάζονται και πώς σχετίζεται, επαναλαμβάνω, η παιδεία με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας των εξτρεμιστικών θέσεων. Ευχαριστούμε πολύ. Ορίστε κύριε Υπουργέ μου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Για να σας απαντήσω λοιπόν, είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο ζητήματα και θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την ε, τρομοκρατία και τα ακραία στοιχεία. Αυτό είχε ζητηθεί, ήταν ε, προαπαιτούμενο δηλαδή για τη συνεργασία με το Πακιστάν και εμείς ε, με τις ίπα προωθήσαμε και της δυνατότητας ανασυγκρότησης στις όμορες περιοχές μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν έτσι ώστε να υπάρχουν ε, επιχειρήσεις, να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα για να μην στρέφεται κάτι, κανείς προς την ε, τρομοκρατία. Παραδείγματο χάρη, ε, οι προτιμησιακές συμφωνίες δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι επλήγησαν και μιλάμε και για ένα κόστος ε, της τάξης των 70 δις. Και υπήρχαν και λιγότερες επενδύσεις ε, εντός του Πακιστάν, γιατί για να γίνουν επενδύσεις θα πρέπει να υπάρχει ένα ασφαλές περιβάλλον. Και τα τελευταία χρόνια δεν εξασφαλιζόταν κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο και δυστυχώς υπήρξαν ε, εισβολές από το Αφγανιστάν στο Πακιστάν και πολλές φαγές στρατιωτών, κάτι το οποίο δεν ε, ενισχύει το οικονομικό περιβάλλον στον ε, κοινωνικό τομέα και στην εκπαίδευση. Σας είπα αρχικά ότι δώσαμε πολλές προσόδους στις ε, περιφέρειες. Και αυτό προβλέπεται και από το Σύνταγμα, δηλαδή η εκπαίδευση είναι δικαίωμα κάθε παιδιού και καθήκον του κράτους να το εξασφαλίζει, να την εξασφαλίζει τα παιδιά. Άρα έχουμε επιτελέσει πρόοδο και είμαστε και ευγνώμονες στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι προώθησε και την προτιμησιακή πρόσβαση στις αγορές και το GSP Plus μας βοήθησε ιδιαίτερα. Γι' αυτό αυτή είναι η καλύτερη εναλλακτική που μπορείτε να προωθήσετε έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην καταφέρουν στην ε, τρομοκρατία. Ο κύριος Charles Τάνοκ έχει το λόγο ως συντονιστής των ε, μεταρρυθμιστών και συντηρητικών και στη συνέχεια έχουμε Σάιετ Μίλαν Μον Σόλτς και Χακ που έχουν ζητήσει το λόγο. Εντάξει, θα σας δώσουμε το λόγο. Αρχίζουμε με τον κύριο Τάνοκ. Ευχαριστώ. Να σας καλωσορίσω και εγώ εξ ονόματος ε, της ομάδας μου που συμπεριλαμβάνει πολλούς ε, συντηρητικούς Βρετανούς και μας ενδιαφέρουν οι εξελίξεις ιδιαίτερα στη χώρα σας. Ε, διαχρονικά έχω, έχω παρακολουθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και εδώ μιλάμε ε, για τα δικαιώματα των μειονοτήτων καθώς και τα εγκλήματα τιμής κατά των γυναικών. Επίσης, εθνότητες ε, που ζουν στο Λονδίνο ε, και βλέπουμε ότι αυτή η διασπορά προωθεί ε, δικά σας ζητήματα. Η μουσουλμάνια Ματία και ο εκπρόσωπος θα βρίσκεται εδώ απόψε. Εμείς γνωρίζουμε ποια ήταν η στάση του έναντι του Πακιστάν και θα θέλαμε να ξέρουμε γιατί αυτή η ειρηνική μειονότητα δεν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά της, ιδιαίτερα στο Μπαγκλαντές. Επίσης, ποια είναι η σχέση σας με την Ινδία μετά την εκτέλεση ε, ενός τρομοκράτη την προηγούμενη εβδομάδα στο Μουμπάι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι σχέσεις θα έχουν μία καλύτερη εξέλιξη μεταξύ Νέου Δελχή και Ισλαμαμπάντ. Εσείς προβάλλετε θέματα άμυνας και τι γίνεται με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, τη δυναμιά Αισαβ; Υπάρχουν στοιχεία, ιδιαίτερα ε, οι μυστικές υπηρεσίες οι οποίες προσπαθούν να δώσουν ιδιαίτερη ίσχυ στους ε, Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Ποια είναι η θέση σας ε, μετά την ISAF ως προς την ενίσχυση των Ταλιμπάν. Μπορούμε να δώσουμε και σε άλλους το λόγο να απαντήσετε στη συνέχεια. Σάιατ. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω, κύριε Υπουργέ, απόψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ είμαι επικεφαλής της ομάδας φίλων του Πακιστάν και θα ήθελα να σας συγχαρώ γιατί σήμερα το απόγευμα είσαστε ιδιαίτερα ε, ακριβείς ως προς την προσέλευσή σας. ως προς το καθεστώς των, ε, πλέ, των ε, πλέον ευνοημένων κρατών που ισχύει στη, για την Ινδία, ζητήσαμε και από την Ινδία και από το Πακιστάν να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και τότε είχε ασχοληθεί ο τότε Υπουργός Εξωτερικών με το θέμα αυτό, σε σχέση με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει και το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο. Ως προς την περίπτωση της ε, Μαλάλα, είναι μια υπόθεση που ε, συγκλώνησε τον κόσμο, όχι μόνο το Πακιστάν. Μιλάμε για κοινέ αξίες που διαθέτουμε, γι' αυτό θεωρήσαμε ότι μπορούσαμε να έχουμε μια κοινή θεώρηση του ζητήματος. Επίσης, τα Αραβικά Εμμυράτα ε, προωθούν το όλο ζήτημα και βεβαίως είναι ευπρόσδεκτη στο Ηνωμένο Βασίλειο και από όσο γνωρίζω έχει ανακτήσει τις δυνάμεις της. Ως προς επικείμενες ε, εκλογές, Υπουργέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει, ε, ε, έχει μάλλον αποστείλει μια ομάδα παρατηρητών, κάτι το οποίο αποτελεί πάγια τακτική μας. Μπορείτε να μας πείτε πώς το, πώς το βλέπετε σε σχέση με αυτή την πάγια τακτική μας. Τέλος, σε σχέση με την πείρα των ε, πολιτών, τις εμπειρίες των πολιτών όταν μεταβαίνουν στο Πακιστάν, δυστυχώς ε, γίνονται ε, πολλές απαγωγές οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και στο σκοτωμό. Είχαμε τρεις περιπτώσεις Βρετανών υπηκόων που σκοτώθηκαν. Κανένας δυστυχώς δεν ε, ήταν υπόλογος. Ο Μαλικ Μαχάλι Ικπακ επίσης πήγε μετέβη στο Πακιστάν για να φέρει πίσω τους υπόδικους και σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε. Επίσης, μια άλλη περίπτωση στο Ηνωμένο Βασίλειο αφορά ένα εξάχρενο κοριτσάκι, την Ατία Άντεμ Βίλκινσον, και από όσοι γνωρίζουμε ο πατέρας της έχει φυλακιστεί διότι ε, την έβγαλε από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ξέρουμε πού βρίσκεται στην επικράτεια του Πακιστάν και θέλουμε να είμαστε σίγουροι από τη δική σας πλευρά ότι δεν αντιμετωπίζει κινδύνους. Θα υποβάλλω το ζήτημα και στο Υπουργείο σας, αλλά θα θέλαμε εσείς να μας εγγυηθείτε ότι θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε τη Βρετανίδα αυτή υπήκο. Συνάδελφοι, Αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Αλλά μακρηγορείτε. Θα ήθελα να είσαστε πολύ πιο σύντομοι. Ο κύριος Μίλαν Μον έχει το λόγο. Ναι. Θα ήθελα ε, να βάλει τα ακουστικά η Υπουργός και θα μιλήσω στην μητρική μου γλώσσα. Εμείς ε, που προερχόμαστε από πιο περιφερειακές ε, χώρες, δυστυχώς δεν μπορούμε να προσέλθουμε με την ίδια ακρίβεια εδώ, όπως είπε ο κύριος ε, Σαλαφράνκα. Μετά την επανεκλογή του Πρόεδρου Ομπάμα, πώς βλέπετε να εξελίσσονται οι σχέσεις των δύο χωρών που κλειδονίστηκαν τα τελευταία χρόνια από όσο γνωρίζουμε. Και βεβαίως είχαν και επιπτώσεις ως προς τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στο Αφγανιστάν και την επανατροφοδοσία τους. Πώς εξελίσσονται οι σχέσεις σας με τις ΗΠΑ και με τον ΝΑΤΟ. Uh, Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ε, η Δευτέρα απόγευμα είναι δύσκολη μέρα για όλα τα, τα κοινοβούλια. Γνωρίζω και από το δικό μας το κοινοβούλιο το τι γίνεται. Κοιτάξτε τώρα, τα τελευταία χρόνια είχαμε δύσκολες ε, σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, και νομίζω πως αυτό φλόταν σε παρεξηγήσεις, γιατί τα σημεία αποκλήσεων τελικά είναι σημεία σύγκλησης, γιατί το Πακιστάν βεβαίως είναι Ε, η χώρα η οποία ενδιαφέρεται περισσότερο για ένα ειρηνικό, σταθερό και Αφγανιστάν το οποίο θα ευημερεί. Και οπωσδήποτε δεν υπάρχει αμφιβολία πως το Πακιστάν θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας επίσης. Γιατί είναι κάτι το οποίο βεβαίω βλάπτει το λαό μας, την οικονομία μας, τη χώρα μας, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Εμείς είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να παλέψουμε οποιαδήποτε ομάδα, ενώ οποιαδήποτε χρησιμοποιεί βία για να ασκήσει πίεση ή για να δείξει τη δύναμή τη. Κατόπιν είπατε το ποιε πρέπει να είναι οι προσδοκίε μας ε, σε σχέση με τον πρόεδρο Ομπάμα. Βλέπουμε ότι στου τελευταίους έξι μήνες ε, έχουμε μια σταδιακή ομαλοποίηση των σχέσεών μα κάτι το οποίο βεβαίω εμπνέει εμπιστοσύνη και δείχνει πω ε, όταν ασχοληθούμε εντατικά με ένα ζήτημα και έχουμε ένα κοινό στόχο, μπορούμε να τα καταφέρουμε και με το Αφγανιστάν και με την περιοχή. Και η προσδοκία μας είναι προφανώς πως το Αφγανιστάν δεν θα υπάρξει κάποιο κενό ασφαλείας ε, και αυτό αναμένουμε από το ΝΑΤΟ, αυτό αναμένουμε από τις ε, ΗΠΑ και οποιαδήποτε άλλη χώρα όμως όσον αφορά τη σχέση μας με τον ΝΑΤΟ, θεωρούμε πως αυτή τη στιγμή έχουμε κοινού στόχους, αλλά θεωρούμε και τη σχέση μας με τον ΝΑΤΟ πάρα πολύ σημαντικές. Ο κ. Σαντάτ Καρύμ αναφέρθηκε στο καθεστώς ε, με την Ινδία. Να σας πω πως στο Πακιστάν το να... με το να αναστρέφουμε μια πολιτική 40 ετών δείχνουμε την επιθυμία μας ε, ε, στο να μεταβάλουμε την κατάσταση με τρόπο ο οποίος θα κοιτάει πλέον το μέλλον και θα κοιτάμε ε, τη σχέση των δύο χωρών από την πλευρά των ε, τοπικών σχέσεων. Γιατί το ξέρετε και στις Βρυξέλλες αναδύονται οι περιφέρειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τις προκλήσεις που έχει είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας ολόκληρης περιοχής η οποία συνεργάζεται και ελπίζουμε και η Νοτιοανατολική Ασία κάποια στιγμή να κάνει το ίδιο και είμαστε υπερήφανοι για αυτό το άνοιγμα προς την Ινδία και ελπίζουμε να βρει ανταπόκριση για την Μαλάλα. Κάνατε ένα σχόλιο, νομίζω πως η κοπέλα αυτή ένωσε το Πακιστάν. Αναφερθήκατε στις εκλογές ε, και στους παρατηρητές. Είναι δουλειά της ε, υπηρεσιακής ε, κυβέρνησης και της Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, αλλά σα διαβεβαιώ πω θα καλωσορίσουμε παρατηρητέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφερθήκατε και σε κάποια άλλα συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν άτομα και ειδικά ζητήσατε να σα δώσω την προσωπική μου άποψη. Οπωσδήποτε θα εξετάσουμε τι λεπτομέρειε τη υπόθεση και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Προ τον κύριο Τσάλ Στάνοκ. Πρώτα απ' όλα, οι πληροφορίες σας πως οι μουσουλμάνοι του δόγματος ε, Αματήρ διώκονται είναι τελείως λανθασμένοι. Ε, ελπίζω να διορθωθεί αυτό, να καταγραφεί στα πρακτικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για οποιαδήποτε μελλοντική συζήτηση. Μάλιστα έχουμε βουλευτές ε, που είναι μουσουλμάνοι Αχματήρ, οπότε δεν απαγορεύεται το δόγμα αυτό μακράν αυτού. Μετά αναφερθήκατε για εγκλήματα τιμή, ε, δολοφονίες γυναικών κτλ. Εγώ παραδέχτηκα ότι το Πακιστάν όπω και άλλε αναπτυσσόμενες χώρε, ε, γύρω γύρω μα, οι γειτονικέ χώρες, δεν ε, έχει έλλειψη προκλήσεων στο πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κοινωνικό κτλ. Αλλά και είμαι η πρώτη που αναγνωρίζω πω τα τελευταία τέσσερα χρόνια το Πακιστάν έχει κάνει μεγάλα βήματα για να αντιμετωπίσει αυτέ τι προκλήσει. και σας έδωσα στην αρχή κάποια παραδείγματα της νομοθεσίας, της προστασίας που δίνουμε στις γυναίκες σε αυτές οι οποίες είναι ευπαθείς οικονομικά, κοινωνικά. Μα η κατάσταση δεν θα αλλάξει από την μια μέρα στην άλλη. Ελπίζουμε η κοινωνία μας ε, να μετασχηματιστεί σε, κάποια, σε, σε μια κοινωνία σαν τις δικές σας. Ναι, αλλά πρέπει να ενθαρρύνουμε βέβαια στον κόσμο για να γίνει κάτι τέτοιο. Μετά αναφέρατε επίσημες ε, κατηγορίες για το δίκτυο Ισάν Αρκανή. Νομίζω πως είναι κάπως ε, καταλειωμένες ε, οι πληροφορίες σας. Η ΙΠΑ εν τω μεταξύ συνεργάζονται με το Πακιστάν και για να σας ενημερώσω πρόσφατα όπως ξέρετε το Κογκρέσο τον είπα, αποφάσισε πως το δίκτυο Χαγκάνη είναι ένα τρομοκρατικό δίκτυο. Εμείς ως χώρα που συνεργαζόμαστε στενά με τις ΙΠΑ ρωτηθήκαμε. Οι απόψεις μας όπως τις μεταφέραμε στις ΙΠΑ και θα ήθελα να τις μεταφέρω και σε εσάς είναι πως δεν έχουμε εμείς δουλειά να εκφέρουμε άποψη για το δίκτυο Χαγκάνη γιατί δεν είναι ε, Είναι αλλοδαποί αν ε, θεωρηθεί ένα τρομοκρατικό δίκτυο, εμείς ευχαρίστως να το κάνουμε. Δεν δίνουμε λοιπόν στήριξη κρυφή ή ανοιχτή σε αυτά τα δίκτυα. Υπάρχει όμως μια πραγματικότητα σε αυτή την περιοχή. Είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και σαφώς έχω πει ε, επανειλημμένος και θέλω να επαναλάβω πως το Πακιστάν θεωρεί για σοβαρούς λόγους πως οποιοδήποτε χρησιμοποιεί βία δεν μπορεί να είναι φίλος του Πακιστάν, κρυφά ή ανοιχτά. Και συνεργαζόμαστε με τους Αφγανούς αδελφούς μας και άλλες φιλικές χώρες για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ένα τον άλλον. Τέλος, με ρωτήσετε κάτι το θέμα, η ερώτηση για τις γυναίκες λοιπά. Νομίζω πως είπατε εκπρόσωπος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Καθιάστον, ε, είναι βεβαίως κάποια η οποία μας κάνει και μας περήφανος και εσείς θα έπρεπε να είστε ε, υπερήφανοι για αυτήν. Είναι και πολύ αποτελεσματική για τα, τις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις θα Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Έχω ακόμη τέσσερα αιτήματα για ερωτήσει Θα λάβετε όλο τον λόγο λοιπόν προτείνω, αλλά βλέπετε πω είναι 4 παρα 10, 4 η ώρα θα έχουμε την ψηφοφορία, οπότε θα σα παρακαλέσω να είστε σύντομοι έτσι ώστε η κυρία Υπουργό να μπορέσει να απαντήσει. Οπότε. Η Μαρίτια Σχάκε, το κ. Χόλτ, Άτκινς και ο κύριος Πόσελτ. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω οι ερωτήσει σα να διατυπωθούν σε ένα λεπτό. Μαρίτιε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι που ανταλλάσσουμε απόψει ε, μαζί σας. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά τις ε, σχέσεις σας με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και πώς το βλέπετε στο γεωπολιτικό πλαίσιο και τις ε, προκλήσεις που εμείς θεωρούμε σοβαρές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο ερώτημα μου αφορά την ελευθερία λόγου και συγκεκριμένα την πρόσβαση σε πληροφορίες στο διαδίκτυο. Ζούμε σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο. Υπάρχουν 50 εκατομμύρια site στο Πακιστάν μόνο. Υπάρχει λοιπόν φιλτράρισμα λογοκρισία σε μια χώρα. Αυτό επηρεάζει και τις άλλες χώρες. Ποια είναι η απόψη. Και επίσης το YouTube εξακολουθεί να είναι απαγορευμένο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί αν ισχύει αυτό και η χώρα σας έχει κάνει κάποια πρόταση στην διεθνή στην ε, συνεδρίαση της ε, Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης που λαμβάνει χώρα στο Ντουμπάι. Έχετε κάποιες προτεραιότητες στον αφορά την κυβέρνηση του Ιντερνετ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σχόλτς. Να ακολουθήσει το καλό παράδειγμα του σεβασμού του χρόνου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς κυρία Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Θα περιοριστώ στο ερώτημά μου και όχι σε γενικότητες. Λοιπόν, πρώτον, ποια είναι η θέση της χώρας σας ως προς την αναγνώριση του καθεστώτος παρατηρητού στον ΟΗΕ της Παλαιστίνης. Δεύτερον και σχετικό, πώς κρίνεται την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Μπανκιμούν να κηρύξει την Παλαιστίνη ως ε, κάποιο είδους ελεύθερη ζώνη εκεί. Και τρίτον ακούμε φήμες για πολύ στενή συνεργασία μεταξύ γερμανικών εργοστασίων όπλων της εταιρείας Κέχλερ Χόχλες με το Πακιστάν που αγοράζει όπλα όπλα που χρησιμοποιούνται παγκοσμίω σε σειράξει και υπάρχουν επίσης φήμες και νέα ότι όπλα που χρησιμοποιούνται ενόμος από αυτή την εταιρεία στη Γερμανία και αγοράζονται στο Πακιστάν χρησιμοποιούνται και στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει δηλαδή εκεί μια σύνδεση που καλό θα ήταν να την ξέρουμε κι εσείς. Και τέλος, ποια είναι η θέση σας για τη διαμάχη στο Κασμίρ. Ευχαριστώ πολύ ο Σερ Άτκινς. Εγώ πάντα είμαι σύντομος πρόεδρε όπως ξέρετε. Ο Ιμπραν Χάν είπε ότι το Πακιστάν είναι από τις πιο διεφθαρμένες χώρες του κόσμου. Αλήθεια είναι αυτό. Και αν ναι πώς το αντιμετωπίζετε. Δεύτερον, ο νόμος για την βλασφημία πότε θα αλλάξει ώστε να μην δολοφονείται κανείς απλώς και μόνο γιατί υπερασπίζεται μη μουσουλμάνους αφού λέτε ότι είναι ελεύθερη χώρα. Ο κύριος Πόσελτ τελευταίος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, έχω δύο κλασικές ερωτήσεις εξωτερικής πολιτικής. Η κυρία Σχάκη αναφέρθηκε στη γεωστρατηγική σημασία του Πακιστάν και θέλω να σα ρωτήσω για τις σχέσεις σας με τις χώρες του κόλπου όπου ζουν πολλοί Πακιστανοί, υπάρχουν παραδοσιακοί δεσμοί αλλά και προβλήματα και βεβαίως μια ερώτηση για την Κεντρική Ασία, Τατζικιστάν, Κυργιζία, το εάν αυτό επιδρά και στο Πακιστάν. Δύο σημαντικές δηλαδή γειτονικέ σας περιοχές. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ. Ευχαριστώ. Νομίζω πως είναι ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις. Και νομίζω πως ε, μας δίνουν έτσι την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε κάποιες παρεξηγήσεις και να αφαιρθούμε βεβαίως σε αυτά τα οποία εμφανίζονται. Κύριε Πόσελτ, αναφερθήκατε στη γεωπολιτική και τη Μέση Ανατολή και το πόσο μας ανησυχούν οι αλλαγές. Νομίζω πως έχουμε στρατηγικές σχέσεις με πολλές χώρες, ειδικά με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου και πολλές άλλες χώρες που υφίστανται μετασχηματισμούς. Εμείς ε, υποστηρίζουμε βεβαίως τις αρχές ελαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας των χωρών και αν υπάρχει ένα εσωτερικό κύμα ε, εντό μιας χώρας ε, που επιθυμεί την αλλαγή, τότε οπωσδήποτε το Πακιστάν το στηρίζει αυτό. Το είδατε στην ε, Αίγυπτο, στην Τινησία. Π.χ. με την Αίγυπτο ελπίζουμε να έχουμε πολύ ισχυρότερε σχέσει από αυτέ που είχαμε με τη μη δημοκρατική Αίγυπτο. Το Πακιστάν είναι δημοκρατική χώρα. Οπότε βεβαίω ε, στηρίζει την ε, αυτόχθονη δημοκρατία όπου εμφανίζεται. Μετά αναφερθήκα στο Τουρκμενιστάν και Τατζικιστάν. Κοιτάξτε, η σταθερότητα οπουδήποτε σήμερα στον κόσμο είναι κάτι το οποίο διασχίζει τα σύνορα και η αστάθεια το ίδιο. Και όσον αφορά αυτές τις χώρες έχουμε καλές σχέσεις ε, μαζί τους και οι δημοκρατία Κεντρικής Ασίας είναι πιο σημαντικές βεβαίως για εμάς γιατί ε, καθώς ελπίζουμε ότι θα σταθεροποιηθεί το Αφγανιστάν θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε ως ε, διαμετακομιστική οδό για να, πάμε τα, να μεταφέρουμε τα προϊόντα μας και να εμπορευτούμε με αυτές τις χώρες. Όπως αναφέρθηκε, στο Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή που μας πέρασε μιλήσαμε για μια εμπορική συμφωνία η οποία θα συμπεριλάβει και το Τατζικιστάν. Συνειδητοποιείτε τι σημαίνει αυτό για το Αφγανιστάν. Θα είμαστε πλέον όλοι συνδεδεμένοι για την σταθερότητα του Αφγανιστάν. Και αν αποτελεί βεβαίω έναν κόμβο διαμετακομιστικό το Αφγανιστάν, θα δημιουργήσει αυτό οικονομικές ευκαιρίες και μια δυναμική δική του. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό για να δοθεί αυτή η ευκαιρία στο Αφγανιστάν. Κύριε Άτκινς, μιλήσατε για τον Ιμραν Χάν και το ότι είπε πως ο Πακιστάν είναι από τις πιο διεφθαρμένες χώρες. Πρώτα απ' όλα, μετά από πολλή δουλειά, τώρα φέρνουμε στο Κοινοβούλιο ιστορική νομοθεσία η οποία θα αφορά τον ελεγχό της διαφθοράς και τη λογοδοσία. Αλλά πιο σημαντικό Θέλω να επισημάνω πως για 3,5 χρόνια η κυβέρνησή μας για πρώτη φορά στην ιστορία του Πακιστάν η Επιτροπή Δημοσίων Λογαριασμών του Κοινοβουλίου είχε ως ηγέτη τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Οπότε αν μια κυβέρνηση ε, ήταν διεφθαρμένη δεν θα έκανε τον ε, επικεφαλή της αντιπολίτευσης πρόεδρο της Επιτροπής Δημοσίων Λογαριασμών. Οπότε έχουμε ένα πρόβλημα όπως και άλλες χώρες με διάφορες μορφές διαφθοράς. Το γνωρίζουμε και είναι μια πρόκληση για το Πακιστάν και γι' αυτό νομοθετούμε ε, για να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αναφέρατε τον νόμο περί βλασφημίας. Ε, να επισημάνω. Και να πω γιατί είναι σημαντική αυτή η ευκαιρία. Από τις 253, δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο, χοντρικά σα τα λέω, 253 υποθέσεις βλασφημίας, μόνο 9 αφορούσαν μη μουσουλμάνους. Όλες οι υπόλοιπες ε, ήταν περιπτώσεις κατά μουσουλμάνων. Οπότε όταν λέτε εργαλείο δίωξης των μη μουσουλμάνων, ε, νομίζω πως ε, είναι μια λανθασμένη αντίληψη. Δεύτερον, κάτι άλλο σημαντικό. Ξέρετε, το να είναι σε διάφορες πρωτεύουσε και το να είμαι εγώ στο Ισλαμαμπάντ και να πηγαίνω συχνά ε, στις ε, πρωτεύουσε, ε, βλέπω και διαβάζω νέα για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πακιστάν. Να σας ρωτήσω το εξή. Ποιος στο Πακιστάν ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Είναι η Daily Telegraph, η New York Times ή όλοι αυτοί λαμβάνουν τις πληροφορίες τους από τον ελεύθερο πακιστανικό τύπο από την κοινωνία των πολιτών του Πακιστάν. Ξέρετε πως όλα αυτά είναι τα, ε, οι οδύνες ε, της γέννησης της πραγματικής δημοκρατίας. Επίσης ε, για τη βλασφημία. Να σας επισημάνω την περίπτωση Ρήμ Σαμασί. Η ίδια κοπέλα η οποία διώχθηκε από κάποιον που έτυχε να είναι χριστιανός ε, διώχθηκε και από έναν μουσουλμάνο. Η ίδια ε, κοινωνία εξέθεσε τον μουσουλμάνο και ε, ο οποίος φυλακίστηκε. Και η κοπέλα τώρα είναι ελεύθερη. Δηλαδή βλέπετε πώς η χώρα και η κοινωνία αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα. Και έχω εμπιστοσύνη πως το Πακιστάν μέσω της κοινωνίας των πολιτών, του Κοινοβουλίου, των ΜΜΕ, αλλά κυρίως μέσω του Κοινοβουλίου και του νομοθετικού έργου που λαμβάνει η χώρα, αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις με ε, τρόπο και προληπτικό. Και ε, γνωρίζουμε πως υπάρχουν αυτές τις προκλήσεις και μας ανησυχούν. Και είναι φυσικό. Απλά επισημαίνω πως γίνονται πολλά. Κατόπιν, μια ερώτηση για το καθεστώς ε, της Παλαιστίνης, ε, το καθεστώς ε, παρατηρητού και βεβαίω υποστηρίζουμε το αποτέλεσμα στον ΟΗΕ και μετά αναφέρθηκε το ότι κατασκευάζονται όπλα υπό άδεια και καταλήγουν κάπου στη Μέση Ανατολή. Εμεί είμαστε μια χώρα η οποία δεν εμπλέκεται σε αυτή τη σύγκρουση που αναφέρατε καθόλου. Πρέπει να πω λοιπόν πως δεν μου ακούγεται πολύ πιστευτό αυτό το οποίο λέτε. Αλλά τι λεπτομέρειες να τις δούμε. Μετά, για το Κασμίρ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εμείς θεωρούμε πως ε, το ζήτημα Τζαμού και Κασμίρ μεταξύ των ε, δύο χωρών ε, έχει επιληθεί. αυτοί οι οποίοι προκαλούν να δημιουργήσουν συγκρούσεις, ε, από ό,τι φαίνεται, δεν θα αφοπλιστούν μέχρι να αντιμετωπιστεί οριστικά το ζήτημα. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Μπορούμε να το λύσουμε με περισσότερες εχθροπραξίες. Το Πακιστάν θεωρεί πως όχι. Μπορούμε να το λύσουμε μέσω πολέμων. Η απάντηση του Πακιστάν είναι όχι. Η απάντηση του Πακιστάν είναι πώς μπορούμε να λύσουμε αυτά τα ζητήματα στην Τράπεζα Διαλόγου. Γι' αυτό πρέπει να συμπεριλάβουμε και ναι. τους δύο εκπροσώπους ε, του λαού του Κασμίρ στο διάλογο για να συνεισφέρουν και αυτοί. Οπότε ερευνούμε και επενδύουμε πάρα πολύ στην, ε, στο διάλογο με την Ινδία για να βρούμε και ξεκινάμε ε, με ζητήματα τα οποία είναι λιγότερα δύσκολα όπως το ζήτημα Σαντζή όπου είχαμε φτάσει κοντά στο να το λύσουμε. Οπότε βεβαίως αυτό μας ε, ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τέλος για την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρεί γεωπολιτική πρόκληση. Ε, Ξεκινώντα την παρέμβασή μου, είπα το ότι η κυβέρνησή μα είναι υπερήφανη για το ότι έχει μια εξωτερική πολιτική που εστιάζεται στην περιοχή και θέλει να βελτιώσει του δεσμού με όλου του γειτονέ μα. Τώρα, Όσο και αν χρειάζεται να βελτιωθούν οι δεσμοί με την Ινδία, το ίδιο πρέπει να γίνει και με το Ιράν, γιατί και το Ιράν την χάνει να έχει σύνορα με το Πακιστάν. Οπότε κάνουμε μια προσπάθεια συνεχή για να βελτιώσουμε τις ε, σχέσεις μας, όπως κάνουμε με όλους τους γειτονές μας. Θεωρούμε πως είναι σημαντικό ε, πως ε, ο μόνος τρόπος σταθερότητας είναι η βελτίωση των σχέσεων Τώρα για το, το πυρηνικό τη πρόγραμμα. Εμείς θεωρούμε πως κάθε χώρα έχει δικαίωμα στην πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτική χρήση και ενθαρρύνουμε το Ιράν να σεβαστεί τι ε, διεθνείς του δεσμεύσει. Μετά για την ελευθερία του λόγου. Ε, πιστέψτε με, εάν έρθετε στο Πακιστάν και δείτε τον τύπο μας θα συμφωνήσετε πως ε, είναι πιο ελεύθερη από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο η ελευθερία λόγου δεν είναι κάτι το οποίο δεν το παίρνουμε στα σοβαρά. συγκεκριμένα για το YouTube και το συμβάν αυτό. Αυτό ήταν αντίδραση σε ε, ένα ζήτημα ασφαλείας που αφορούσε το Πακιστάν και όπως είχε γίνει και σε πολλές άλλες χώρες Block that one particular... Ζητήσαμε το YouTube να μπλοκάρει το συγκεκριμένο site, το οποίο δεν μπόρεσαν να κάνουν και άρα αναγκαστήκαμε να μπλοκάρουμε το YouTube. Μόλις συμφωνήσουμε να μπλοκάρουν συγκεκριμένα site που δημιουργούν ε, προβλήματα και ανησυχίες, ευχαρίστως ε, να το ξεμπλοκάρουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Υπουργέ για την παρουσία σας και για το ότι άμεσα δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να απαντήσετε στα ερωτήματά μας. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Ε, ζητώ συγγνώμη για τις καιρικέ συνθήκες. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Thank you. Thank Γεια σας συνάδελφοι, αρχίζουμε με τις ψηφοφορίες ε, γιατί έχουμε μεγάλη μερίσια διάταξη. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι μετά θα συζητήσουμε για την κατάσταση στην Αίγυπτο. ευχαριστώ κύριο Μπερναρντίνο Λεόν, ο οποίος είναι ο ε, και υπεύθυνο για θέματα Νότιας Μεσογείου. Ε, αυτό το πρώτο θέμα θα πρέπει να το ε, ψηφίσουμε για δεύτερη φορά. Εταιρική κοινωνική ευθύνη, πρόθεση συμφερόντων της κοινωνίας και πορεία προς μια βιώσιμη ανάκαμψη. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Amendment 1 in favor. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, με συγχωρείτε, μαζί με την προφορική Υπαριθμό ένα με την προφορική. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ. Α, όχι, όχι, καταπίπτει, με συγχωρείτε. Τρία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προφορική δύο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4. Καταπίπτει συμβασμός 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβασμός 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σαράντα ένα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σαράντα δύο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σαράντα τρία υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω θα πρέπει να ελέγξουμε την 43. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 45 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι 46 ηλεκτρονική επαλήθευση ένας λείπει πέρας απορρίπτεται rejected to it. Uh, Απορρίπτεται. 19 υπέρ και 27 κατά. Τώρα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το σχέδιο γνωμοδότησης. Παρακαλώ ψηφίστε. One more colleague. Λείπει ένας. Εντάξει, φαίνεται ότι δεν θα ψηφίσει. Πέρας. Εγκρίνεται με 41 ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά. Η κυρία Ντάτη. Πρόεδρε. Ασάιφη, όχι Ντάτη, ναι. υπερψήφισα και φάνηκε σαν να έχω απόσχη. Ναι. Λάθος, λάθος. Okay. we need to vote again on Ψηφίζουμε λοιπόν για τη γνωμοδότηση αυτή και αρχίζουμε με την τροπολογία 1. Κύριε Μάουρο, έχετε το λόγο επειδή πρέπει να ξαναψηφίσουμε τα ίδια, εάν συμφωνούν ε, οι ομάδες να κρατήσουμε τον κατάλογο ψηφοφοριών, ας ε, ψηφίσουμε μόνο το τελικό σχέδιο. Αφού πρέπει να ψηφίσουμε δύο φορές. Εάν έχουν όλες οι ομάδες ε, όλες τον ίδιο κατάλογο και συμφωνήσουν γι' αυτό. Αντιτίθεται κανείς. Στην τροπολογία 40 είχε προσθεθεί μια προφορική και την πρώτη φορά δεν την ψηφίσαμε. Τώρα που είναι δεύτερη, ίσως να την ψηφίσουμε. Πώς 40, αλλά με την προφορική 5 δεν εκπίπτει, όχι γιατί αν καταψηφιστεί απλώς θα ισχύσει η 39. Η γραμματεία ίσως ξέρει καλύτερα. Η προφορική τροπολογία 5 καταπίπτει αν εγκριθεί η συμβιβαστική 10. Έτσι μου λέει η γραμματεία. Εδώ γράφει αν εγκριθεί και αν εγκριθεί και η συμβιβαστική 10 τότε θα συμπεριληφθεί στο κείμενο της τροπολογίας 40 ως προσθήκη. Ως προσθήκη. Α, δηλαδή κάναμε λάθος που δεν ψηφίσαμε για την προφορική 5. Αυτό εννοείται. Αυτό μας λέτε δηλαδή. Ίσως να έχετε και δίκιο. Ναι, ναι, μάλλον, αλλά να είναι δύσκολα εδώ. Ναι, συνάδελφοι, αν δεν έχετε αντίρρηση να ψηφίσουμε την προφορική 5 πρώτα και μετά όπως ζήτησαν οι ομάδες να μην ξαναψηφίσουμε δεύτερη φορά. Λοιπόν, προφορική 5. Περ. Α, πρώτα ο εισηγητής. Κοιτάξτε, κοιτάξτε είμαι κατά της τροπολογίας αυτής, διότι υποτίθεται ότι συμπεριλαμβανόταν στον συμβιβασμό, αλλά την Παρασκευή το απόγευμα, Παρασκευή το απόγευμα, είμαι λοιπόν κατά. Είμαι κατά της προσθήκης. Είστε κατά. Α, δηλαδή δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε τότε. Δεν μπορούμε. και θα πάμε στο επόμενο. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, με συγχωρείτε. Λοιπόν, όπως είχαμε συμφωνήσει οι πολιτικές ομάδες, δεν θα ξαναψηφίσουμε τώρα. Θα κρατήσουμε τα αποτελέσματα της πρώτης ψηφοφορίας. Συνεχίζουμε με το επόμενο θέμα του κυρίου Μάουρο. Ως προς την συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράκ. Ας αρχίσουμε λοιπόν 56 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ ε. κατά αποχές θα πρέπει να ελέγξουμε συνάδελφοι 64 ελέγχουμε ηλεκτρονικά Please uh, show the results. Close the vote. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεν ήταν σαφής θέση των σοσιαλιστών. 65 που είναι ίδια με την 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 75 και 80 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77-79 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτονται. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σύμβασμος 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ όχι με συγχωρείτε 101 κάτσιν υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 101 Πέρας. Απορρίπτεται. Με δύο ψήφους διαφορά. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112-113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 115 με την προφορική 1 η κυρία Κοπά θα ήθελα να προτείνω μια προφορική που θα είχε ως εξής αναγνωρίζει τις συνεχείς δεσμεύσεις των αρχών του Ιράκ έτσι ώστε ε, οι κάτοικοι των καταβλισμών να διαβιούν υπό ε, κανονικές συνθήκες και μέσα στα πλαίσια της ε, διαδικασίας συνεργασίας θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τον επαναπατρισμό των κατοίκων του καταβλισμού φαρία έτσι ώστε να διευθετηθεί το όλο ζήτημα της επανεγκατάστασης ή επαναπατρισμού. Ο κύριος Μάουρο. Πρόεδρε, θα αντιταχθώ σε αυτή την προφορική γιατί στην πρόταση, την προφορική που έχει υποβληθεί, υπάρχει η επαναπατρισμου ο κυριος μαουρο θα αντιταχθω σε αυτη την προφορικη γιατι στην προταση την προφορικη που εχει υποβληθει υπαρχει η δυνατοτητα ε, ε του ζητήματος μέσα στα πλαίσια του καταβλισμού αυτού και θεωρώ ότι θα πρέπει να μην περιπλέξουμε τα πράγματα ως προς τη συνέχεια της ψηφοφορίας. Άρα αντιτάσσεστε στην προφορική. Ναι, κατά της προφορικής των σοσιαλιστών. Η κυρία Κοπά. Και εμείς... Κατά της προφορικής τροπολογίας του ΕΛΚΑ. Οπότε δεν θα ψηφίσουμε καμία προφορική τροπολογία και ψηφίζουμε την 115 χωρίς προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές δεκτή η 115 η αρχική, χωρίς την προφορική τροπολογία. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 119 να την επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται με δύο ψήφους. Διαφορά. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να την επαληθεύσουμε και αυτή. η Ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της 120. Close the Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψηφοδιαφορά. 122. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 128 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 129 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 130 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 131 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 132 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 6 στο εκτιμώντας α υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 19 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 21 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 22, 25 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή Τροπολογία 33 με προφορική τροπολογία 2. Κύριος Κασίν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να υποβάλω μια προφορική τροπολογία ε, ως συμβασμό που έχει ως εξής. Ενώ ένα γραφείο στο Ερμπίλ θα μπορούσε να... Εκτιμώντας ότι ένα γραφείο στο Ερμπίλ θα μπορούσε να αυξήσει την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ. Γιατί πολλές εταιρείε έχουν ε, γραφεία στο Ερμπίλ και όχι στη Βαγδάτη. Και όλοι πάνε εκεί πέρα οι επιχειρηματίε. Γι' αυτό νομίζω πως με την τροπολογία αυτή μπορούμε να βοηθήσουμε το γραφείο μας να είναι εκεί, να έχει ε, ορατότητα και να στηρίξει τις δραστηριότητες στο Ερμπίλ. Ευχαριστώ. Είναι κάποιος κατά. Ψηφίζουμε λοιπόν. την τροπολογία 33 με την προφορική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές. Δεν είναι σαφές. Ε, επαληθεύσουμε την τροπολογία 33 με την προφορική τροπολογία 2 του κ. Κατσίν. Πέρας. Απορρίπτεται Περνάμε στην 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στη 41. Εάν δεν έχει κανείς αντίρρηση, από την 41 έως την 50 όλες μαζί. Πλην 43 ε, λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Και τώρα η τροπολογία 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως εγκρίνεται αν θέλετε να την επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται και αυτή. 52 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 54. Στην 54 θα πάμε γιατί 30 δεν πέρασε. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και 55 επίσης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται περνάμε στα, σε σκέψει σκέψεις από 1 έως 14 ε, μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτές όλες Θα ψηφίσουμε τώρα ηλεκτρονικά στο σύνολο. Okay, please close the vote. Πέρας της ε, ψηφοφορίας εγκρίνεται 49 υπέρ 2 αποχές.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 Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου γνωμοδότησε στην ε, ΑΦΕΤ θεωρώντας ότι θα πρέπει να επιτευχθεί η συνένεση και έχουμε μια τελική ψηφοφορία ψηφίζουμε υπέρ ή κατά ηλεκτρονικά. Τελική ψηφοφορία. Oh, sorry, sorry, No. Again, we need to repeat again. Sorry, there was a technical. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία. Ανέκυψε ένα τεχνικό πρόβλημα. Λείπουν τρεις. Two more? One more? <laughs> Τρεις, δύο, ένας. Okay, let's close the vote. It's adopted... Uh... Εγκρίνεται. Με 47 ψήφους υπέρ και δύο αποχές. ένταξη μεταναστών, συνέπειε στην αγορά εργασίας και συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης. Έκθεση Βαν Πρέντα. Προφορική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ, κατά

46 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και μία αποχή. Ο κύριος Πρέντα ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Κάναμε λάθος όταν ψηφίσαμε το δεύτερο τμήμα της 2 γιατί ε, εγκρίθηκε η προφορική τροπολογία υπαριθμών 1 είχα μια ξεχωριστή ψηφοφορία στη 2 και δεν χρειαζόταν να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα διότι είχε εγκριθεί η προφορική υπαριθμών 1. Έχετε δίκιο. Αλλά είχε νομίζω έτσι κι αλλιώς ε, απορριφθεί το δεύτερο τμήμα, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, το καταγράφουμε. Ευχαριστώ. So that was the last uh, dossier for the... Τελευταίο θέμα ψηφοφορίας και θα συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, την ε, κατάσταση στην Αίγυπτο, αλλά έχουμε λίγα λεπτά διάλειμμα πριν. Colleagues, I just learned that Mr. Leon will be here at 5 o'clock. That means we have an interruption. Θα διακόψουμε για 20 λεπτά περίπου. 15 με 20. Ξαναρχίζουμε στις 5. Προσπαθούμε να βρούμε και να φέρουμε τον κύριο Λεόν το συντομότερο δυνατόν. Υπότιτλοι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 So, colleagues, we can uh, ναι, Αδελφοί, ξεκινάμε και ο κύριος Λέων ήρθε. Το επόμενο θέμα λοιπόν είναι η Αίγυπτος. Καλώς ορίζω τον κύριο Περναρδίνο Λεόν, ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της ε, Μεσογείου και υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την δήλωση της 22ης ε, Νοεμβρίου του Πρόεδρου Μόρση που βεβαίως είναι αντιβαίνει στους, στον έλεγχο και στη διάκριση των εξουσιών στο κράτος δικαίου καθώς δίνει ασυλία σε όλες τις προεδρικές αποφάσεις και στην έκδοση διαταγμάτων. Ε, κάτι το πολύ ανησυχητικό. Η συνταγματική αυτή δήλωση η οποία προστατεύει το ε, Συμβούλιο την Σούρα δηλαδή και την συντακτική συνέλευση από διάλυση εκδόθηκε εν αναμονή της απόφασης του ανώτατου συνταγματικού δικαστηρίου για το θέμα. Οι συνταγματικές αυτές δηλώσεις έρχονται σε μια στιγμή κρίσιμη για την δημοκρατική διαδικασία στην Αίγυπτο όπου θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συζητούν το σχέδιο συντάγματος εν ώψη του δημοψηφίσματος το Σύνταγμα της 15ης ε, Δεκεμβρίου και εκλογές ε, στις ε, το 2013. Βεβαίω, διάφοροι εκπρόσωποι μεταξύ των οποίων και εσεί τονίσατε ξανά την μεγάλη σημασία των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στην Αίγυπτο καθώ και την κεντρική σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για μακροπρόθεσμη οικονομική βοήθεια στην Αίγυπτο και στηρίζει την Αίγυπτο στις προσπάθειές της για να ανακάμψει από το καθεστώς Μουμπάρακ. Στις ε, ανταλλαγή απόψεων μαζί σας σήμερα θα θέλαμε να συζητήσουμε ποια οικονομικά και πολιτικά μέσα έχουν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πιέσει την Αίγυπτο για να, ε, τηρήσει, να διατηρήσει το κράτος δικαίου, το διαχωρισμό και τον έλεγχο των εξουσιών καθώς επίσης ε, και βλέπουμε πως αυτό είναι μια σημαντική δοκιμασία για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία και τι αντίκτυπο μπορεί να έχει η αρχή περισσότερα για περισσότερα, τι μοχλούς έχει για να πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ε, ανάκτηση διαφόρων περιουσιακών στοιχείων. Επίσης θα πρέπει... Clear about the foundation of... Πρέπει να είμαστε επίσης σαφείς για την βάση της σχέσης αυτής, δηλαδή σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών ελευθεριών και μια ανεκτική κοινωνία στο πλαίσιο του κράτους δικαίου. Κύριε Λεόν, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας δώσω τον λόγο για να ακούσουμε τις παρατηρήσεις σας και τις σκέψεις σας και μετά θα έχουμε τη δυνατότητα για να ακούσουμε τις παρεμβάσεις των συναδέλφων και τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Με μεγάλη χαρά επιστρέφω στο Κοινοβούλιο. Σήμερα συζητούμε την Αίγυπτο που ξέρω ότι σας ενδιαφέρει όλους πόσο μάλλον που τις τελευταίες δύο εβδομάδες είδαμε ότι αυξάνουν οι πολιτικές διαφωνίες μεταξύ των τριών παραγόντων του πολιτικού τριγώνου, δηλαδή τον πρόεδρο και τη μουσουλμανική αδελφότητα με το κόμμα της που, στηρίζουν και που το στηρίζουν και ορισμένα άλλα κόμματα, το δικαστικό κλάδο και τα αντιπολιτευόμενα κόμματα. Αυτές οι διαφορές ε, χειροτερεύουν από τη δήλωση της 22ης Νοεμβρίου Οπότε και η Σούρα δήλωσε ο πρόεδρος ότι πρέπει να έχει ασυλία κατά προσφυγής από το συνταγματικό δικαστήριο. Μετά το σχέδιο συντάγματος εγκρίθηκε με πολλές διαφωνίες όπως ξέρετε. Το πρωί της Παρασκευής 30 Νοεμβρίου και μετά την έγκριση του συντάγματος ανακοινώθηκαν διαδηλώσεις από μη μουσουλμάνους την Παρασκευή και από μουσουλμάνους το Σάββατο. Και εκεί εμφανίστηκαν ακόμη περισσότερες εντάσεις στο Κάιρο και αλλού. Πολλές εντάσεις όχι βέβαια ακραία βία, αλλά πολλές εντάσεις. Ο πρόεδρος Μόρση ζήτησε δημοψήφισμα για το Σύνταγμα στις 15 Δεκεμβρίου. Τέλος το ανώτατο δικαστήριο, το συνταγματικό δικαστήριο, αναμενόταν να αποφανθεί χθες για τη Σούρα και τη Συμβουλευτική Συνέλευση, αλλά οι Ισλαμιστές περικύκλωσαν το κτίριο και διαδήλωσαν. Και το κόμμα ελευθερίας και δικαιοσύνης, δηλαδή το κόμμα των μουσουλμάνων αδελφών, ζήτησε να μην εμποδιστεί το έργο των δικαστών. Τελικά το δικαστήριο αποφάσισε να παγώσει τις συνεδριάσεις του μέχρι νεοτέρας διαταγής. Ξέρετε ότι έχει ζητηθεί από τους δικαστάς να μποϊκοτάρουν το δημοψήφισμα. Αργά την Κυριακή οι δικαστές ανακοίνωσαν ότι αρνούνται προς στιγμή να συμβιβαστούν και επαναλαμβάνουν την θέλησή τους να μην επιτηρήσουν στο εξής τις εκλογές αν και η απόφαση αυτή δεν είναι δεσμευτική για όλα τα μέλη του δικαστικού. Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο κατηγορήθηκε ότι παρεμβαίνει σε πολιτικά θέματα και το Εθνικό Μέτωπο Σωτηρίας καταδίκασε την έκκληση του Μόρση για δημοψήφισμα. Σημαντικές δε πολιτικές προσωπικότητες όπως ο Άμρ Μούσα έκαναν δηλώσεις που έλεγαν ότι το σχέδιο συντάγματος ε, υποβλήθηκε πολύ γρήγορα και δεν μπόρεσε ο κόσμος να το συζητήσει. Πολλά πολιτικά κόμματα εξέφρασαν ανάλογες απόψεις και ανακοίνωσαν για αύριο διαδηλώσεις και συλλαλητήρια μπροστά στο Προεδρικό στο Κάιρο. Μια δήλωση υπογράφτηκε από 18 πολιτικά κόμματα και οργανώσεις καθώς και το Συνταγματικό Κόμμα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το Εθνικό Μέτωπο Δικαιοσύνης και Ελευθερίας, η κίνημα της 6ης Απριλίου και το κίνημα Κεφάγια. Η αντιπολίτευση είτε μποϊκοτάρει το δημοψήφισμα είτε προτείνει αρνητική ψήφος αυτό. Αλλά δεν συμφωνούν όλες οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις ούτε οι συμπολιτευόμενες. Ακούγονται και φωνές που προτείνουν άλλες λύσεις. Πριν από μερική ώρα Ακούστηκε νέα πρόταση από τον, από τον πρώην πρόεδρο του Οργάνωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που προτείνει να βρεθούν μερικοί συμβιβασμοί για συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολιτευτικών δυνάμεων η πάτη εκπρόσωπος και η ίδια η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων καθώς και εγώ ο ίδιος είμαστε σε συνεχή επαφή με τους σημαντικότερους παλιτικούς παράγοντες τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Πρόεδρο, εκπροσώπους από τα περισσότερα κόμματα, από την κοινωνία των πολιτών και τους λέμε πάντα ότι το θέμα είναι να υπάρξει μια συνένεση μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων για να υπάρξει συμφωνία με τον δικαστικό τομέα και να αποφευχθεί έτσι η θεσμική διαμάχη και να ξανασυνεχίσει η συζήτηση του συντάγματος με όλους τους τομείς της κοινωνίας με σεβασμό της ένομης τάξης και του ανεξάρτητου δικαστικού κλάδου. Με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας κλπ. Αυτά μάλιστα τις βασικές δημοκρατικές αυτές αρχές τις επαναλαμβάνουμε συνεχώς σε όλους τους Αιγυπτίους συνομιλητές μας και συνομιλήτριες γιατί θέλουμε να οικοδομηθεί μια σωστή δημοκρατία με σεβασμό του αχωρισμού των εξουσιών και όλα αυτά με σεβασμό και των μειονατήτων. Μπορεί να είδατε την πρόσφατη μου δήλωση όπου έλεγα ότι ο σεβασμός των μειονατήτων είναι ένα κλειδί της δημοκρατίας, δεν αφορά μόνο τις εκλογές, αλλά είναι γενικότερη αρχή στην πορεία της μετάβασης και φυσικά η ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα, η ελευθεροτυπία, η ελευθερία της έκφρασης, όλα αυτά είναι μας. Από αυτή την άποψη λοιπόν ήμασταν σαφείς. Κάθε πλευρά έχει τα επιχειρήματά της, αλλά το σημαντικό για μας είναι να επιμείνουμε στην εξέβρεση συνενέσεων Πιστεύουμε ότι το Προεδρικό Διάταγμα δεν έτυχε τέτοια συνένεση και ήταν λάθος άρα. Και πιστεύουμε επίσης ότι η οικοδόμηση τέτοια συνένεση είναι ευθύνη όλων των Αιγυπτιακών πολιτικών δυνάμεων και όλων των πολιτικών παραγόντων. Βεβαίω ειδικότερη ευθύνη έχει η κυβέρνηση, ο πρόεδρος, αλλά είναι πάντως ευθύνη όλων των πολιτικών παραγόντων. Μάλιστα πρόσφατα, όπως υπενθύμησε και ο πρόεδρος, υπάρχει αυτή η Task Force Αιγύπτου Ένωσης που είναι εξαιρετικό εργαλείο που διαθέτουμε για να συνεργαστούμε με τους Αιγυπτίους και τις Αιγύπτιες. Δεν είναι αυτός σκοπός βέβαια, δεν είναι, είναι απλώς η αρχή μιας διαδικασίας συνεννόησης με τη Ένωσης και Αιγύπτου. Οι συνεργάτες μας έχουν ορίσει αυτή τη σχέση ως ένα νέο συμβόλαιο με την Αίγυπτο. Και το λέμε αυτό στην τελική μας δήλωση για την προώθηση της σταθερότητας, της ειρήνης, της συγνωνικής δικαιοσύνης, της ευταξίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της καλής διακυβέρνησης, governance. Είναι πολύ καλό εγγραφό αυτό. Και οι παράγραφοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, τη συνένεση είναι πάρα πολύ στεναρά διατυπωμένες. Και υπάρχει και το θέμα της μεγάλης υποστήριξης των Ευρωβουλευτών. Μερικοί από αυτούς είναι παρόντες σήμερα, ο κύριος Σαλαφράγκα, ο κύριος Ότεμπροκ, όλα αυτά, όλα αυτά είναι σημαντικά. Έχουμε επαφές και με προσώπους της κοινωνίας των πολιτών και στις συνεδριάσεις και μετά και πριν τις συνεδριάσεις των μελών της Task Force. Συναντιόμαστε με προσώπους πολιτικών κομμάτων, αντιπολιτευομένων κομμάτων, για να υπάρχει και πλουραλισμός. Και έτσι ανοίγουμε νέους δρόμους για τον διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών και θεσμών των δύο πλευρών. Μπροστά μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε ανήφορο. Οι προσεχείς εβδομάδες μέχρι το δημοψήφισμα αλλά και μετά από αυτό δεν θα είναι εύκολες. Αλλά πιστεύουμε στεναρά ότι η απάντηση πρέπει να είναι περισσότερη Ευρώπη στην Αίγυπτο. Δηλαδή περισσότερη δουλειά της Ευρώπης στην Αίγυπτο για να μπορέσει να συμβάλλει στη δημιουργία αυτής της συνένεσης. Αυτή είναι η απάντηση. Είναι η Ένωση ο μόνος διεθνής παράγοντας που θα ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο εργαλείο όπως αυτήν την Task Force και την τελική αυτής δήλωση. Και λόγω της μοναδικής αυτής θέσης και των ευθυνών που έχουμε, φαίνεται ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε, δηλαδή να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με όλους τους γεφυροποιούς. Think. Δεν θα είναι εύκολο βέβαια, γιατί και η Υπηρεσία των Εξωτερικών Δράσεων αλλά και οι Ευρωβουλευτέ μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο και τους ενθαρρύνουμε να τον παίξουν αυτόν τον ρόλο με τους συνομιλητάς τους στην Αίγυπτο. Η συνεννόηση με τις κυβερνητικές δυνάμεις, με αντιπολιτευόμενες δυνάμεις, με θεσμικά όργανα στην Αίγυπτο, διότι, διότι η λύση για την Αίγυπτο είναι κάτι που θα ωφελήσει τους πάντες και την Ένωση και ολοκλήρη την περιοχή. Επιμένω λοιπόν. Περισσότερη Ευρώπη, περισσότερο ρόλο στην Αίγυπτο, περισσότερη δέσμευση και στενή συνεργασία με όλους όσους προσπαθούν να οικοδομήσουν γέφυρες. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε κύριε Λεόν. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στα μέλη που μετέβησαν στην Task Force στο Κάιρο, ε, Σαλαφράγκα και Νέτς. Ο κύριος Σαλαφράγκα έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω και τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αίγυπτο και για τη θέση που διατύπωσε στην, στο διευρυμένο Προεδρείο αυτής της Επιτροπής για την ανησυχητική κατάσταση που ε, ζουν οι Αιγύπτιοι γιατί μετά την ε, αίσια έκβαση της Task Force στην Αίγυπτο είδαμε ποιες ήταν οι εξελίξεις. Θα ήθελα να αναφέρω στον κύριο Λεόν ότι είχαμε την εντύπωση μαζί με την κυρία Νέης στην Επιτροπή ΣΟΥΡ. Θεωρήσαμε ότι είχαν προχωρήσει οι εργασίες και έπρεπε λοιπόν να δούμε κατά πόσο η Σαρία θα είναι η βασική πηγή που θα διέπει το νέο σύνταγμα. Αυτό που μας είπαν οι εκπρόσωποι μειοψηφιών ήταν ότι προσπαθούν να φτάσουν σε μία συνένεση, αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε. Η ύπατη εκπρόσωπος κατέβαλε μια προσπάθεια επί του θέματος, αλλά δυστυχώς δεν είχε έκβαση το ζήτημα. Ποια θα ήταν λοιπόν η εναλλακτική αν το συνταγματικό δικαστήριο που ακύρωσε ήδη την Βουλή θα είχε ακυρώσει και την συντακτική συνέλευση και ποια είναι η εναλλακτική που έχουμε ενώπιον μας. Δηλαδή τι θα γίνει ε, ως προς το σύνταγμα το οποίο ορίζει την, ε, τις εκτελεστικές εξουσίες και τα καθήκοντα του Πρόεδρου Μόρση για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ποια θα ήταν λοιπόν η εναλλακτική λύση ε, σε, στην περίπτωση που δεν ε, εγκριθεί το Σύνταγμα. Και ποια είναι η αξιολόγηση της ΕΙΕΔ του συντακτικού κειμένου που δεν βασίζεται σε δημοκρατικές αρχές αλλά σε μια μειοψηφία και πώς θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε μια συνένεση με βάση μια νέα πρόταση. Τέλος, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο πιστεύετε ότι με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες, εάν δεν αρθεί αυτό το διάταγμα, όπως πιστεύουν μερικοί, αλλά εγώ έχω ορισμένες επιφυλάξεις, θα πρέπει να αρθεί και η αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ επί του θέματος, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι είπα συνδράμουν στρατιωτικά αυτή τη χώρα. Ε, ευχαριστούμε κύριε Σάρλα Φράγκα. Η κυρία Νέης το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, εξ ονόματος της ομάδας μου, να ευχαριστήσω τον κύριο Λεόν που ήρθε εδώ και είναι έτοιμος να συζητήσει ένα θέμα πολύ δύσκολο και μια κατάσταση επίσης ε, Κανθόδη. Εγώ ήμουν μία από τις ε, ευρωβουλευτές ε, που συμμετείχαν στην ομάδα που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Από τη μία βεβαίως με εντυπωσίασαν οι απαντήσεις που έλαβα από ομολόγους μας της Σούρας και τους μουσιογράφους. Δηλαδή μας έλεγαν αυτά που ήξεραν ότι θέλαμε να ακούσουμε. Αυτή ήταν η εντύπωση που είχα, αλλά σκέφτηκα εντάξει, ο καιρός θα δείξει. Ο χρόνος θα δείξει. αν θα κάνουν αυτά που λένε ή αν είναι μόνο λόγια. Αυτό ήταν το ένα. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση ε, σε μια τρίωρη συζήτηση που είχαμε με μέλη της Σούρας από τρία κόμματα είναι όχι η παράνοια, η σχεδόν παράνοια ναι. που τους διακρίνει η απόρριψη δηλαδή οποιασδήποτε ενέργειας θα μπορούσε να φανεί ως ε, παρέμβαση από το εξωτερικό. Το τρίτον που πρέπει να θυμόμαστε positive role είναι ο ρόλος που έπαιξε ο πρόεδρος Μόρση στην ε, ο διαμεσολαβητικός του ρόλος για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Δεν μπορούμε έτσι να το ξεπεράσουμε έτσι απλά. Είναι πολύ σημαντικό και τέλος, πριν από λίγα χρόνια, σκεπτόμενοι, έπρεπε να το έχουμε πει αυτό στο ε, παρελθόν. Δηλαδή τα λάθη που έγιναν μετά τον πρώτο γύρο των ελεύθερων δημοτικών εκλογών στην Αλγερία που βγήκαν οι Ισλαμιστές και ο δεύτερος γύρος δεν έγινε ποτέ. Και υπήρξε μια ανακούφιση ανά τον πλανήτη σχεδόν και μετά τι έγινε, τι είχαμε χάος και εμφύλιο πόλεμο στην Αλγερία. Αυτά πρέπει να τα έχουμε κατά νου του των λεχθέντων. Πρέπει να ομολογήσω πως αισθάνομαι τουλάχιστον αμηχανία από το ότι ο πρόεδρος Μόρση, αφού ήταν συμπρόεδρος σε μία από τις συνεδριάσεις ε, της ε, Task Force και μας μίλησε για τη δέσμευσή του στη δημοκρατία, μετά από λίγες μέρες εξέδωσε το γνωστό διάταγμα, ε, το οποίο κανείς μας δεν εγκρίνει. Αυτό το οποίο πρέπει να αναρωτηθούμε λοιπόν είναι ποια είναι η ενδεδειγμένη πορεία έτσι ώστε τα, αυτά, τα διατάγματα αυτά να ανακληθούν ε, είτε να τροποποιηθούν. Θα γίνει αυτό με δημόσια επίπληξη του Προέδρου ή υπάρχουν άλλοι τρόποι. Και τελευταία ερώτηση προς τον κύριο Λέων. Θεωρείτε πως ε, εάν δεν πάει πολύ άσχημα το δημοψήφισμα ε, θα έχουμε τροποποιήσεις του διατάγματος ε, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση ή θεωρείτε πως δεν υπάρχει καμία ελπίδα και θεωρείτε πως ο καιρός της πίεσης ε, του νέου και έφραυστου παρελθόντος έχει ήδη φτάσει. Ευχαριστώ κυρία Νέιτς. Να δώσω τον λόγο στον κύριο Παντσέρη, πρόεδρο της Αντιπροσωπής για το Μαγκρέμπ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν αμφισβητώ το γεγονός ότι ο πρόεδρος Αιγύπτου διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο για την ανακοχή και γι' αυτό έτυχε και διεθνούς αναγνώρισης. Αυτή η αναγνώριση όμως χρησιμοποιήθηκε από τον Μόρση για να προβάλλει μία ε, στεναρά στάση που οδήγησε στους ε, κλειδονισμούς αυτού στη χώρα. Το Μεσανατολικό είναι ένα ζήτημα χωρίς ε, πάτο. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο αυτές οι ταραχές αποτελούν μέρος ε, μια στρατηγικής για να εξέβρει κανείς νέους χώρους δράσης. η Αιγυπτιακή κοινωνία αντιμετωπίζει νέα γεγονότα και εκβάσεις που εμείς ε, δεν μπορούμε να κρίνουμε απόλυτα. Πρόκειται για μία εσωτερική σύγκρουση. Συμφωνώ με τον Σαλαφράγκα που αναφέρει ότι θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε ως προς το κείμενο του συντάγματος ναι. κάθε αυτού κατά πόσο δηλαδή ανοίγουμε, διανοίγουμε επικίνδυνες οδούς. Δεν νομίζω ότι αρκεί να πούμε ότι είμαστε διαθέσιμοι και είμαστε παρόντες. Θα πρέπει να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να μιλήσουμε για την αρχή του more for more μέσα στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας. Επίσης, ως προς το ρόλο των ΙΠΑ, αναρωτιέμαι πώς εντάσσεται εδώ, ιδιαίτερα ως προς τις στρατιωτικές δυνάμεις και στρατιωτικές ενισχύσεις γιατί έχω την εντύπωση ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Ευχαριστούμε κύριε Παντσέρη. Η κυρία Κιλνέρσεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Λεόν για αυτή την ενδιαφέρουσα εισήγηση, καθώς και τους συναδέλφους που παρέστησαν στο Κάιρο σε αυτή τη συνάντηση. Σύμφωνα με αυτά που είπε και η κυρία Νέης. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει μετά την ανακοίνωση αυτού του διατάγματος ε, από τον πρόεδρο Μόρση. Ο κύριος Αλαφράνκα μίλησε για επιτυχία της Task Force. Όμως οι μη κυβερνητικέ εξέφρασαν την απογοήτευσή τους. Αναφέρουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ότι δεν ε, μπόρεσαν να συμμετάσχουν σε αυτό το σχήμα, δηλαδή δεν δέχτηκε την παρουσία του ο Μόρση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι δέχτηκε αυτή τη θέση του Προέδρου Μόρση. Θα ήθελα να επαληθεύσω αυτή την πληροφορία, κάτι το οποίο μπορεί να κάνει ο κύριος Λεόν και αναρωτιέμαι κατά πόσο αυτή τι η βασική θέση ως προς τις ε, ΜΚΟ και την ε, κοινωνία των πολιτών δεν ενθάρρυνε τον κύριο Μόρση, δεν τον εξώθησε στο να λάβει τις μεταγενέστερες αποφάσεις. Θα ήθελα τυχόν επιβεβαίωση, γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο αποδυναμώνεται η θέση μας ενώπιον του Πρόεδρου Μόρση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Νίλσεν. Όπως αναμενόταν έχουν ζητήσει πολύ το λόγο. Παρακαλώ λοιπόν οι συνάδελφοι να περιορίσουν τις παρεμβάσεις τους σε δύο λεπτά. Θα γίνουν δύο γύροι ερώτα απαντήσεων. Λέω δύο ακόμη. Κυρία Σάκε πρώτη. Δύο-δύο να γίνονται οι ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Λεόν. Μας μιλήσατε για τη σημασία που έχει ο ρόλος που μπορεί να παίξει η Ένωση στην Αίγυπτο η οποία μπορεί να καταστεί υπόδειγμα μετάβασης στη δημοκρατία αλλά αντιμετωπίζει τρομερές προκλήσεις. Είδαμε μεγάλο ενδιαφέρον τι μας είπε η ύπατη εκπρόσωπος μετά την ε, κατάληψη θα έλεγα της εξουσίας από τον πρόεδρο Μόρση. Διάβασα ό,τι έγραψαν οι δημοσιογράφοι και υπήρχε και μια δήλωση για την ανάκτηση ορισμένων χρημάτων από την Αίγυπτο. Για γενικότερη όμως στρατηγική για την Αίγυπτο και τις χώρες της Βορείου Αφρικής θεωρείται ότι καλύπτεται από την ιδέα more for more. Και η Πάτη εκπρόσωπος είπε ότι εδώ είναι η πραγματική δοκιμή, αν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να πράξουμε αυτά που λέμε. Ορισμένοι συνάδελφοι, γιατί κάναμε συζητήσεις, αναρωτήθηκαν μήπως δεν πρόκειται για μια επικίνδυνη στιγμή άμα να λέμε τέτοια λόγια εγώ πιστεύω ότι η υπόσχεση που δώσαμε στον Αιγυπτιακό λαό ότι θα τονίσουμε ιδιαίτερα τις ελευθερίες και τα δικαιώματά τους είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι η στιγμή να δείξουμε ότι η δημοκρατία είναι κάτι παραπάνω από το καθένας μία ψήφο. Γιατί υπάρχει το θέμα της κατανομής των εξουσιών και των ελέγχων. Πόσο σοβαρή θα είναι η Ένωση λοιπόν θα φανεί τώρα αν βάλει όρους για την οικονομική βοήθεια. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την Αίγυπτο, αλλά για ολόκληρη τη στρατηγική more for more. Πότε θα μιλήσουμε λοιπόν επιτέλους για αυτούς τους όρους που πρέπει να βάλουμε. Και τέλος, ποιος είναι ο κύριος συνομιλητής μας, οι κυβερνήσεις ή οι λαοί. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε απλώς αν δεν επικαλεστείτε τώρα την αρχή more for more, πότε θα το πράξετε. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα η κυρία Μουνίθ για δύο λεπτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λεόν για την παρουσία του και θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη δημιουργία της Task Force γιατί αποτελεί ένα μέσο διαλόγου με την κοινωνία των ε, πολιτών για να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε, να διορθώσουμε μάλλον τα λάθη του παρελθόντος που διαπράξαμε στην Αίγυπτο. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε αυτή τη συνένεση όπως αποτολμάει η ΑΕΕ και θα πρέπει να αντιταχθούμε στο ρεύμα που επικρατεί και να δούμε τι θα κάνουμε ως προς την οικονομική αρρωγή. Νομίζω ότι θα φτάσουμε στο σημείο εκκίνησης εάν δεν επανορθωθεί το θέμα του συντάγματος. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λεόν κατά πόσο αλλάζει η θέση της Αιγύπτου τώρα με την αναγνώριση της Παλαιστίνης αναγνώριση ως ε, παρατηρητή στον ΟΗΕ και κατά πόσο αυτό αλλάζει τον συσχετισμό δυνάμεων και με την Αίγυπτο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λέων έχει το λόγο τώρα για να απαντήσει σε αυτό το πρώτο γύρο ερωτήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στον κύριο Σαλαφράν κάποια θα ήταν η εναλλακτική θα είναι δύσκολο να φανταστούμε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Αλλά όχι, το φανταστούμε πως χωρίς το διάταγμα και την αναστολή του χτες από το συνταγματικό δικαστήριο την, η Ισούρα και η συντακτική συνέλευση θα χρειάζονταν ένα χρόνο για να ξαναδούν όλα τα κείμενα, το σχέδιο συντάγματος κτλ. Οπότε όλοι εμείς σήμερα θα ασκούσαμε κριτική στην απόφαση αυτή, εάν είχε ληφθεί στην Αίγυπτο. Αυτό το οποίο όμως είναι σίγουρο, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, είναι πως έχουμε μια κατάσταση στην οποία όλες οι πιθανές επιλογές είναι κακές. Σαφώς. Και όλες οι πλευρές έχουν κάποια επιχειρήματα. Και, και θετικά και αρνητικά. Και σωστά και λαθασμένα και από πλευράς ουσίας, δημοκρατίας δηλαδή και οικοδόμησης της δημοκρατίας και από τις σκοπιά της διαδικασίας δηλαδή συνένεσης και συμπερίληψης ως τα μέσα της μετάβασης αυτής. Οπότε, τώρα έχουμε αυτό το σύνταγμα το οποίο έχει εγκριθεί. Νομίζω πως ε, από λίγο καιρό. Βεβαίως θα έχουμε νέες ε, συναντήσεις με τους εκπροσώπους της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης ή με εμένα και θα μπορέσουμε να δούμε το σύνταγμα αυτό σε περισσότερη λεπτομέρεια. Αλλά η πρώτη αξιολόγηση δεν αφορά τόσο το τι υπάρχει στο σύνταγμα, αλλά το τι δεν υπάρχει. Το κείμενο καθε αυτό προσπαθεί να παραμείνει σχετικά ουδέτερο Υπάρχουν κάποια σημαντικά ζητήματα που λείπουν. Δικαιώματα γυναικών δεν υπάρχουν στο κείμενο. Αλλά νομίζω πως χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να αξιολογήσουμε το Σύνταγμα και έχουν εντύπωση πως δεν έχουμε χρόνο να μπούμε σε λεπτομέρειες. θα μπορούσε, όπως είπατε και εσείς και άλλοι, η κυρία Σχάκη είπε, Mr. Panseri, should we uh, cancel uh, our support to Egypt? Μήπως λοιπόν πρέπει να ακυρώσουμε την ε, βοήθειά μας προς την Αίγυπτο. Να ξεκαθαρίσω πρώτα απ' όλα πως έχουμε συμφωνήσει σε κάποια προγράμματα πλαίσιο. Πως ο, η στήριξή μας πάντοτε ε, είναι υπό την, την, αίρεση, την διαφόρων όρων και βεβαίω τη αρχή περισσότερα για περισσότερα. Αυτά είναι ξεκάθαρα, το έχει πει ο Επιτροπός Φίλε στις ανακοινώσεις του Μαρτίου και του Μαΐου Οπότε όλα τα προγράμματα που έχουμε συμφωνήσει είναι οι παρτές της αιρέσεις και δεν μπορώ τώρα να δώσω μια απάντηση για το τώρα ή σε δύο εβδομάδες ή σε έξι μήνες γιατί πάντα, συνέχεια, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε αυτές τις δύο αρχές τούτων λεχθέντων. Οπότε πρέπει να αξιολογήσουμε την κατάσταση και ε, πώς θα οδηγηθούμε ίσως σε ένα πάγωμα, πιθανό πάγωμα της βοήθειας προς την Αίγυπτο. Κοιτάξτε, ε, λίγο πριν έρθουμε εδώ πέρα, λάβαμε κάποιες προτάσεις, η τελευταία ήταν από τον ε, Αλσαντάτ. Και καθώς έχουμε αυτή την ε, μοναδική θέση και η κυρία Νέιτσο Αουτεμπρούκ το είχε δει αυτό όταν ήταν στο Κάιρο πριν από λίγες εβδομάδες. Έχουμε λοιπόν αυτή τη μοναδική θέση και πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία λοιπόν ε, λαμβάνομαι μια θέση απεμπλοκή θα ήταν πλήγμα αυτό για τους Αιγυπτίους που προσπαθούν να βρουν μια λύση. Ρωτήσατε για τις ΕΙΠΑ και, και ο κ. Φαντσέρη το ρώτησε. Ε, είμαστε σε στενή επαφή με την Αμερικανική Πρεσβεία, τις Αμερικανικές ομάδες που ασχολούνται με την Αίγυπτο και νομίζω πως έχουμε παρόμοιες θέσεις Θέλουμε να επανέλθει λοιπόν αυτή η συνένεση. Και νομίζω πως η κυρία Νέιτς τον είπε κάτι πολύ σημαντικό. Οι Αιγύπτιοι πάντα, αλλά ειδικά τώρα, ανησυχούν για τυχόν παρεμβάσεις. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ διπλωματικοί Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι λιγότερο ελκυστικό ίσως από πλευράς ε, δήλωσης αρχών, αλλά πιο ρεαλιστικό. Αλλά το να μιλάμε ξεκάθαρα και με ειλικρίνεια με τους ε, συνομιλητές μας είναι πολύ σημαντικό και όπως είπα η κυβέρνηση έκανε λάθος ε, στον τρόπο έγκρισης ε, του διατάγματος και στο ότι δεν αναζήτησαν συνένεση και το ξεκαθαρίσαμε αυτό στους συμβούλους του Πρόεδρου. Ε, ρωτήσατε κυρία Νίλσεν κατά πόσο έχουμε αποκλείσει ΜΚΟ. Όχι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν θα μπορούσαμε βεβαίως να καλέσουμε και όλες τις ΜΚΟ ε, που δρούν στην Αίγυπτο. Έπρεπε να κάνουμε μία επιλογή για να έχουμε μία σωστή εκπροσώπηση και είναι γεγονός ότι ορισμένες οργανώσεις δεν ε, κλήθηκαν αλλά καλέσαμε όλους όσους έδρασαν και επικριτικά ως προς το καθεστώς. Δεν μπορούσαμε να καλέσουμε τους ε, πάντες βεβαίως. Έγινε μια πρώτη συνάντηση πριν από την ε, Task Force με τον ειδικό ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπου ακούσαμε γνώμες και ανησυχίες μετά συναντηθήκαμε με εκπροσώπους της κοινωνίας ε, των πολιτών μαζί με τον Επίτροπο Φούλε. Είχαμε περίπου 40-50 μήκυο που συμμετείχαν σε αυτό το σχήμα. Ήταν ένα αρκετά ευρύ σχήμα και στη συνέχεια στο δείπνο μας εκπροσώπησε ο Επίτροπος Φίλε καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της, είχα καθώς και εκπρόσωποι της κοινωνίας των ε, πολιτών. Ήταν ένα πολύ ευρύ σχήμα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αποκλεισμοί. Δεν ε, είχαν ε, κληθεί πάντες και στις τρεις αυτές συναντήσεις, αλλά είναι μία απαρχή της διαδικασίας. Άρα θα ισχύσει αυτό το σχήμα μη αποκλεισμών και αν συνάδελφοι δικοί σας έχουν υποδείξεις ή επαφές ΜΚΟ που έχουν αποκλειστεί και θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην επόμενη Task Force, με μεγάλη χαρά να τους δεχτούμε. Νομίζω ότι απάντησα στην ερώτησή σας. Θα πρέπει πάντα να ορίζουμε τα ζητήματα που αφορούν αρχές. Αυτό το αναφέρω και στην κυρία η ιδιαίτερα. Βεβαίως η λέξη συνένεση είναι η λέξη κλειδί. Και η Γάζα και το παλαινιστινιακό ζήτημα διαδραματίζει και αυτό το ρόλο του. Και ο πρόεδρος Μόρση θεώρησε ότι ήταν αρκετά δυνατός ώστε να προβάλλει αυτό το διάταγμα χωρίς να προβεί σε διαβουλεύσεις. Δηλαδή θεωρούσε ότι η θέση του είναι ακλόνητη. Ευχαριστούμε κύριε Λέοντα. Δεύτερος γύρος τώρα. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λεόν γιατί άμεσα ανταποκρίθηκε στην ε, πρόσκλησή μας και νομίζω ότι θα πρέπει ε, καταρχήν να πω ότι είναι λυπηρό, λυπηρές οι εξελίξεις στην Αίγυπτο τις δύο τελευταίες ε, εβδομάδες και δεν νομίζω ότι ε, μια task force η οποία ήταν επιτυχής ε, θα μπορούσε να επιλύσει και τα πάντα βεβαίως. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα κοινά προγράμματα, τα κοινά συμπεράσματα πρόκειται για ε, θέματα που είχαν ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο και νομίζω ότι 5 δις, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα πέντε δις που υποσχεθήκαμε για τα επόμενα χρόνια. Λυπηρό βεβαίως το, το γεγονός αυτών των εξελίξεων και ο κύριος Λεόν μιλά για συνένεση, αλλά δεν ξέρω, επειδή η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα ταραχώδης, πώς θα μπορούσαμε να προβάλλουμε κάτι τέτοιο. Δεν θα μπορούσε να επιληθεί το ζήτημα ούτε με ένα δημοψήφισμα μετά από την πόλωση των πολιτικών τάσεων και ομάδων. Και δεν νομίζω ότι ε, σε 16 μέρες μπορούμε να προβούμε στην άρση αυτής της πόλωσης της πολιτικής κατάστασης και δεν υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις. Δεν υπάρχει μαγική λύση. Η κατάσταση είναι άκρος ανησυχητική και δεν νομίζω ότι το περισσότερο Ευρώπη επιλύει τα θέματα των Αιγυπτίων. Γιατί η αρχή του μη παρεμβατισμού είναι ιερή αρχή. Εάν το διάταγμα αυτό αρθεί, δηλαδή αν εγκριθεί το σύνταγμα, γιατί έτσι κατάλαβα από το τύπο, αυτό που έχει σημασία όπως και να έχει είναι η πόλωση η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε ένα δεκαπενθήμερο. Η κυρία Ρομέρο από την αντιπροσωπεία του Μαγκρέμπα, αλλά μόνο για δύο λεπτά παρακαλώ ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Λεόν για την εργασία του στη δύσκολη αυτή μετάβαση της Αιγύπτου. Και συσχετίζοντας το θέμα αυτό με το προηγούμενο, θα ήθελα να σας πω τι προβλέπετε αν παγιωθεί αυτή η κατάσταση υπάρχουν περιθώρια εξέβρεσης συνένεσης και τι θα γίνει σε σχέση με έναν απότερο νικητή από αυτή τη διαδικασία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Μόρση ακολούθησε στάση ισχυρού άνδρα και είναι πολύ δύσκολο αυτή η Προεδρία να μπορέσει να ανταποκριθεί και αυτό ισχύει και σε άλλες χώρες της Βορείου Αφρικής. Ποιο εναλλακτικό σενάριο θα μπορούσαμε να προβάλλουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άτκινς για δύο λεπτά. Ε, πρόεδρε, μήπως ε, έχουμε πλέον ε, στιγματιστεί από την εγκύτητά μας με τον κύριο Μόρση και το ότι λέτε ότι πρέπει να εμπλακούμε ακόμη περισσότερο είναι λανθασμένο. Δεν ξέρουμε πώς θα κλείσουν τα πράγματα. Κατόπιν δεν μας είπατε τίποτα για τον στρατό. Εγώ υποτίθεται πως θα πήγαινα στην Γάζα προσφάτως ε, και με σταμάτησαν γιατί υπήρχαν προβλήματα στο Βόρειο Σινά. Αν μπορείτε λίγο να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί. Και τέλος και το Αλτζαζίρα και το BBC μεταδίδουν πως οι δικαστές είναι διχασμένοι για το συνταγματικό δημοψήφισμα. Κάποιοι εμπλέκονται, κάποιοι όχι. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει. Ευχαριστώ, κύριε Άτκινς. Τον κύριο έχει ο κύριος Πόσελτ για δύο λεπτά. Ναι κύριε Πρόεδρε, ανησυχώ για την Αίγυπτο, αλλά καμιά φορά ανησυχώ και για τον ρεαλισμό μας. Ζητάμε από αυτές τις χώρες, δικαίως, να είναι λαϊκές και δημοκρατικές χώρες. Μα το να είναι λαϊκό κράτος ε, είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται απ' έξω σε αυτές τις χώρες ε, και δεν σημαίνει περισσότερο περισσότερη δημοκρατία, ίσως σημαίνει περισσότερο Ισλάμ. Επίση δεν ξέρω εάν εμείς εκπροσωπούμε την πλειοψηφία του Αιγυπτιακού λαού ε, ενώπιον του Προέδρου. Μην ξεχνάμε επίσης πως είχαμε εδώ πέρα και την ε, Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν που εκφράστηκε πολύ θετικά. Πριν από 14 μέρες είχαμε Τουρκούς πολιτικούς στο Στρασβούργο που μίλησαν πάρα πολύ θετικά. Οι Παλαιστίνοι αναφέρθηκαν ήδη και πρέπει να πω πως ο πρόεδρος Μόρση είναι ένα υπόδειγμα θα έλεγα για ολόκληρη την περιοχή Δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο εμείς θέλουμε και υποθέτουμε. Για να είμαι ξεκάθαρος, εγώ θεωρώ πως τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμια και είμαι υπέρ της δημοκρατίας και πρέπει να εμπλακούμε, αλλά μην έχουμε ψευδεστήσεις. Και θα ήθελα να ρωτήσω, με εντάξεις, για ευρωπαϊκές χώρες έχουμε ξεκάθαρα κριτήρια. Τα κριτήρια της Κοπενχάγης, αλλά ποια είναι τα κριτήριά μας στην πολιτική της γειτονίας. Τα έχουμε διατυπώσει, είναι ρεαλιστικά Ευχαριστούμε κύριε Πόσελτ. Και τώρα τον λόγο έχει κυρία Ο κύριος Γιάννης με συγχωρείτε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί πολλά προελέχθησαν τα οποία με βρίσκουν σύμφωνο. Ιδιαίτερα αυτά που, είπε κυρία, που είπαν οι κυρίες Μουνίθ και Ρομέρο έθεσαν το θέμα πώς θα το έθετα και εγώ. Όπως είπε και ο εκπρόσωπός μας, ο κύριος Λεόν. Πιστεύω ακράδαντα στη συνένεση και στο διάλογο και πολλές φορές φτάνουμε σε ανέλπιστα αποτελέσματα μέσω του διαλόγου. Και κάτι που δεν είπε ο κύριος Λεόν πριν από τη συνένεση, υπάρχει οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Και αυτό δεν σημαίνει ότι κάνουμε έκκληση σε καλή θέληση, αλλά θα πρέπει μέσω της ε, διπλωματικούς, ε, διπλωματικής οδού να ε, παραχωρήσουμε και στα συμβαλόμενα μέρη αυτό που επιθυμούν. Αυτά που επιθυμούν. Γιατί δεν υπάρχει μαύρο και άσπρο. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις ενδιάμεσες που διέπουν και την παρούσα κατάσταση. και η ύπατη εκπρόσωπος ε, καθώς και η ΕΔ και εμείς δεν θα έπρεπε να σπεύσετε στις κυρώσεις, κάτι το οποίο δεν θα ήταν ιδιαίτερα ευεργετικό στην παρούσα φάση. Ευχαριστούμε κύριε Γιάννης. Ο κύριος Λεόν έχει το λόγο για να απαντήσει στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν τον κύριο Μιγιάννη. Δεν είναι κρίμα αυτό που είπατε, αντίθετα. η Task Force μας έχει δώσει ένα εργαλείο για να παίξουμε μεγαλύτερο ρόλο στην Αίγυπτο. γιατί έτσι μπορούμε να δουλέψουμε αντιμετωπίζοντας μακροπρόθεσμες προκλήσεις που δεν αφορούν μόνο τον τωρινό πρόεδρο αλλά ολόκληρη την Αίγυπτο αλλά και για τους Ευρωπαίους. Πρέπει να προετοιμάσουμε το έδαφος γιατί δημιουργία θέσεων απασχόλησης πολύ σημαντικό για την Αίγυπτο και δεν αφορά αυτή την κυβέρνηση αυτόν τον πρόεδρο. Είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας και στο μέλλον. Επίσης η Task Force που αντιμετωπίζει επομένως αυτές τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Ήταν επίκαιρη η δημιουργία της χρειαζόταν αυτό το εργαλείο και ό,τι αποφάσισε θα εφαρμοστεί με βάση τις αρχές του more for more. Και το, οι Αιγύπτιοι οι συνομιλητές μας τώρα ξέρουν με το εργαλείο αυτό τι να αναμένουν, αλλά επίσης και πώς να το πετύχουν ή τι δεν μπορούν να πετύχουν. Έτσι είναι τα πράγματα πιο σαφή. Τώρα, πώς να επιτευχθεί η συνένεση. Είπα και πριν ότι ακούστηκαν προτάσεις τον κύριο τη λέει ο και θα ακουστούν και άλλες σύντομα μερικές θα μιλήσουν για προσωρινή έγκριση ή του υπάρχοντος σχεδίου συντάγματος ή κάποιου τροποποιημένου. Άλλες προτάσεις λένε ότι μπορεί να χρειαστούν ορισμένες τροποποιήσεις αλλά που τώρα είναι ακόμη πολύ φλού. Αυτό είναι προτιμότερο αντί να πούμε εμείς τους Αιγύπτιους τι πρέπει να κάνουν γιατί όπως λέει πάντοτε και η πάτη εκπρόσωπος αυτό είναι αιγυπτιακό θέμα και ο δικός μας ρόλος είναι απλώς να τους στηρίξουμε. Αλλά εκείνοι θα βρουν τη λύση. Το διάταγμα, για να απαντήσω και προς την κυρία Ρομέρο, ή μάλλον το τι θα γίνει αν εγκριθεί το σχέδιο συντάγματος. Ο πρόεδρος μας λέει ότι προσπαθεί να μην παρατείνει αυτήν την κατάσταση εκτάκτων εξουσιών που έχει ο πρόεδρος. Μόλις εγκριθεί το Σύνταγμα προβλέπει μία ρήτρα ότι οι νομοθετικές εξουσίες αμέσως θα δοθούν στη Σούρα στο, στη Βουλή. Και αμέσως θα κληθούν νομοβουλευτικές εκλογές και τότε το Κοινοβούλιο θα ανακτήσει τις προσωρινές αυτές εξουσίες που έχει ο Πρόεδρος. Αλλά ρώτησε επίσης η κυρία Ρομέρο τι θα γίνει αν εγκριθεί το Σύνταγμα. Κοιτάξτε, εμείς προβλέπουμε πολύ μικρή διαφορά μεταξύ του ναι και του όχι. Ας δούμε όμως πώς θα τοποθετηθούν οι διάφορες πολιτικές δυνάμεις για το δημοψήφισμα και πώς θα αντιδράσουν μετά τα αποτελέσματα. Προς τον κύριο Άτικιν, η δέσμευση της Ένωσης και της υπάτης εκπροσώπου δεν αφορά ποτέ ένα πρόσωπο, είτε τον πρόεδρο είτε ένα κόμμα, αλλά με ολόκληρη την Αιγυπτιακή Δημοκρατία. Αρνηθήκαμε επανειλημμένως να οργανώσουμε την Task Force προηγουμένως γιατί δεν υπήρχαν οι συνθήκες. Αν και κατανοούσαμε, όπως και η υπόλοιπη διεθνή κοινότητα, ότι οικονομικά η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη στην Αίγυπτο. Αλλά με το ρόλο που έπαιζε ο στρατός μέχρι πρόσφατα δεν νομίζαμε ότι υπήρχαν οι δημοκρατικές συνθήκες που απαιτούνταν για να δημιουργηθεί. Και, και το Δουνουτού συνεφώνησε πρόσφατα με την Αίγυπτο, η ΙΠΑ επεξεργάζονται συμφωνία και άλλοι διεθνείς παράγοντες επίσης και κανείς από μας δεν συνομιλεί με συγκεκριμένο πρόσωπο ή κόμμα, αλλά με την Αιγυπτιακή Δημοκρατία. Ρωτήσατε για το στρατό. Ο στρατός παρέμεινε σιωπηλός στην κρίση αυτή. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Αν δηλαδή αποφάσισαν να αλλάξουν ρόλο όπως ζήτησε ο πρόεδρος Μόρση, δεν εξέφρασαν πάντως, από ό,τι γνωρίζω, καμία συγκεκριμένη θέση για αυτή την κρίση, για αυτά τα προβλήματα. Το Σύνταγμα, ένα από τα στοιχεία του, θα μπορούσε να είναι ο ρόλος του στρατού. Παραδείγματος χάρη το άρθρο εκείνο όπου έχει το δικαίωμα ένα στρατοδικείο να δικάσει πολίτες. Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ δικαστικών, ναι υπάρχει. Δεν συμφωνούν όλοι οι δικαστές. Μερικοί θεωρούνται από τους Αιγυπτίους συνομιλητές μας ως πολύ κοντινοί στο καθεστώς Μουμπάρακ. Άλλοι δε είναι πλήρως ανεξάρτητοι και θέλουν να επιμείνουν στην ανεξαρτησία αυτή. Είναι λοιπόν χωρισμένοι, όπως και πολλοί άλλοι στην ομάδα του πληθυσμού, αλλά δεν μπορώ να σας πω πόσοι είναι υπέρ ποιου. Θα το μάθουμε σε λίγο. Για τον κύριο Πόσελτ τώρα συμφωνώ, συμφωνώ και το έχουμε πει και στα συμπεράσματα της Task Force ότι είναι καθολικά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι είναι σημαντική η Αίγυπτος ως πρότυπο για την περιοχή της και άμα διαβάσετε τα συμπεράσματα, δεν τα έχω μπροστά μου τώρα αλλά θα σας τα στείλω, θα δείτε πόσες φορές μιλάμε για την αρχή αυτή της καθολικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα δείτε επίσης ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία δεν για το πώς βλέπει η Ένωση τα πράγματα. Η Task Force δημιουργώντας αυτό το μεικτό όργανο όπου συμφώνησαν και οι Αιγύπτιοι για τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία μας, τα είπε ρητά. Και τέλος, για τον κύριο Γιάννη σωστά τα είπε. Το θέμα είναι να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη και δυστυχώς αυτό ακόμα λείπει. Θα θέλαμε οι διάφοροι παράγοντες να επιδεικνύουν περισσότερη εμπιστοσύνη μεταξύ τους και ελπίζουμε ότι θα προσπαθήσουν να το κάνουν. Μας λένε ότι γνωρίζουν, ότι έχουν συνείδηση ότι χρειάζεται περισσότερη συνένεση. Και εμείς τους λέμε μην προσπαθείτε τόσο να επαναλαμβάνετε ο καθένα τις θέσεις σας, αλλά περισσότερο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνη και για την εξέβρεση κοινού εδάφους. Συμφωνώ επίσης μαζί σας ότι προς στιγμή δεν είναι ώρα για ακυρώσεις. Ας αξιολογήσουμε πρώτα την κατάσταση, να περιμένουμε μερικές εβδομάδες και μετά η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων της Ένωσης σε συνεννόηση με άλλα κράτη-μέλη κλπ. θα δει τι άλλες επιλογές υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις. Ανοιχτή διαδικασία θα είναι αυτή, όλα παίζουν. Αλλά να περιμένουμε μέχρι την κατάλληλη στιγμή. Σας κατευχαριστούμε κύριε Λέοντα για την παρουσία σας σήμερα. Σας ευχόμαστε επιτυχία. Πριν λήξουμε το θέμα αυτό θα ήθελα να μιλήσει ο κύριος Ιβραήμ Λαχύρ. Μας πει δυο λογάκια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή παρακολουθεί τα πρόσφατα γεγονότα στην Αίγυπτο και έχουμε διαβουλεύσει σε τακτά χρονικά διαστήματα με την ΕΙΕΔ και με τον ειδικό αντιπρόσωπο στην περιοχή. Ασχοληθήκαμε με την προετοιμασία της Task Force κατά την διοργάνωση καθώς και τα συμπεράσματα και χαρήκαμε με την έκβαση της Task Force με, το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου. Όπως είπε και ο κύριος ε, Λεόν, αυτό είναι η απαρχή μιας νέας διαδικασίας συνεργασίας με την Αιγυπτό. Συμφωνώ με τον κύριο Λεόν για τους κανόνες που ισχύουν για την άρση των μέτρων αρρωγής, η κατάργησή τους, που βασίζονται σε συγκεκριμένες αξίες και στην αρχή του more for more, όπως αναφέρθηκε στις δύο περσινές ανακοινώσεις. Εργαζόμαστε υπέρ του Αιγυπτιακού λαού το 2012 δημιουργήσαμε νέες θέσεις εργασίας στις φτωχότερες περιοχές της Αιγύπτου και προωθήσαμε εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης. Το νέο χρήμα που θα μπει στην Αίγυπτο θα ακολουθήσει στην αρχή More for More και παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση. Ευχαριστούμε κύριε Λαφία και με την παρέμβαση αυτή κλείνει το θέμα της Αιγύπτου. Ευχαριστούμε κύριε Λεόν, σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. We are going with the next point of our agenda. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερησία διάταξη, έκθεση πρόοδου 2012 για τη Σερβία έχουμε την πρώτη εξέταση του σχεδίου αυτού έκθεσης. Έχουμε επίσης ε, και το σχέδιο έκθεσης του κοσφοπεδίου δεδομένων των στενών σχέσεων της στενής ε, σύνδεσης των δύο χωρών και βεβαίως ε, είχαμε ταξιδέψει και στο κοσφοπέδιο μετά την δημοσίευση της εκθέσης Κομισιόν και πριν δημοσιευτεί η έκθεση της ε, Επιτροπής αφού ε, πήγαν οι βουλευτές Βελιγράδη και Πριστίνα και βεβαίως ε, ακούσαμε και είχαμε και τον κύριο Βιγγένιν που ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπής. Θα δώσω τον λόγο τώρα στον κύριο Κατσίν, τον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι αυτή είναι μία από τις πιο θετικές εκθέσεις για την Σερβία τα τελευταία έξι χρόνια που ήμουν εισηγητής ε, για την χώρα. Ε, είχα κάνει κάτι ανάλογο και για το Μαυροβούνιο. Παρά τι προκλήσει, λοιπόν, η Σερβία έχει κάνει σημαντικά βήματα τελευταία προ σωστή κατεύθυνση. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο σχέδιο έκθεση παρά το ότι έπρεπε να είναι σύντομη γιατί υπάρχει ένα όριο 6.000 λέξεων και δεν μπορούμε έτσι να κάνουμε θαύματα. Πάνω απ' όλα θα ήθελα να καλωσορίσω την πρόοδο της ε, Σερβίας ε, στις σχέσεις με το Κοσμοπέδιο. Ο διάλογος υψηλού επίπεδου έχει ξεκινήσει. Είχαμε μια ιστορική συνάντηση μεταξύ των Πρωθυπουργών. Ή βρίσκονται σήμερα στις Βρυξέλλες, ε, σήμερα και αύριο, τρίτη φορά τον τελευταίο μήνα η εφαρμογή της Συμφωνίας για Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων θα ξεκινήσει σε μία εβδομάδα από σήμερα. Η δε ε, συμμετοχή της κυβέρνησης του Κωσφοπεδίου στα τοπικά φόρα έχει καταργήσει την αυτοαπομόνωση της σερβικής κυβέρνησης. Αλλά Βελιγράδη και Πριστίνα δεν έχουν κάνει πραγματικό διάλογο εδώ και 25 χρόνια. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια και βεβαίως μια σταθερή ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Και βεβαίω η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει ένα ρόλο κλειδί. Ταυτόχρονα η Σερβία αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση στην καταπολέμηση τη συστημική διαφθορά και του οργανωμένου εγκλήματο. Δράτω με τη ευκαιρία να καλωσορίσω τι προσπάθειε του κυρίου Βούτσιτς, αντιπροέδρου της κυβερνήσεως. Πρέπει να εθαρρύνουμε την κυβέρνηση να συνεχίσει αυτή την πορεία. Η κυβέρνηση, η έκθεση με συγχωρείτε, τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης ε, των mm. μεγάλων περιπτώσεων διαφθοράς. Οι δημόσιες προμήθειες ε, mm. και η εμπλοκή των ιδιωτικών συμφερόντων παραμένουν πηγή διαφθορά. Επίση, ενθαρρύνουμε τι ελληνικέ αρχέ για να συνεχίσουν με τι μεταρρυθμίσει. Ο κύριο Βούτσιτ επίση γνωρίζει πώ θα συναντηθεί με του εκπροσώπου Σέρβων που ζουν νότια του ποταμού Ήμπαρ που είχαν αγνοηθεί εντελώ μέχρι στιγμή από το Βελιγράδι. Καλωσορίζω αυτέ τι ανακοινώσει και ελπίζω η συνάντηση αυτή να λάβει χώρα σύντομα. Οπωσδήποτε πριν το τέλο του έτου. Από την άλλη, τονίζεται στο σχέδιο έκθεση η ανάγκη διατήρησης της ανεξαρτησίας ε, των θεσμικών οργάνων του κράτους, ε, καθώς είχαμε αλλαγή του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας με την ανάληψη καθηκόντων της νέας κυβέρνησης. Επιπλέον, είχαμε την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης που αντιμετώπισε πολλά προβλήματα το περασμένο έτος. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και ο επαγγελματισμός δικαστών και εισαγγελέων και να αποκατασταθεί η πίστη των πολιτών στη δικαιοσύνη. Η ανάκαμψη της ερβικής οικονομίας ε, και η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σχετίζονται άμεσα με την πρόκληση αυτή. Η έκθεση θα ασχοληθεί ειδικά με το ζήτημα του ποινικού κώδικα, οι διατάξει του οποίου έχουν βεβαίως συχνά παραβιαστεί από εισαγγελείς ε, και επίσης έχουν αποτελέσει αντικείμενο κατάχρησης όπως το άρθρο 359. Θα παρακολουθούμε λεπτομέρεια τις εξελίξεις για την εφαρμογή των συστάσεων μας. Επίσης, δυστυχώς σημειώνουμε πως το Pride Parade απαγορεύτηκε φέτος στο Βελιγράδι. Ένα κρίσιμη, μια κρίσιμη δοκιμασία για την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων είναι να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα μεταξύ των οποίων και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ. Η ελευθερία έκφρασης ε, έχει κορυφαία σημασία σε όλες τις ευρωπαϊκές ε, δημοκρατίες και στην Σερβία. Τέλος, θεωρώ πως πρέπει να αναφερθώ στις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την περίπτωση ε, των κρατών στρατηγών και του Ραμούς Χαραντινάη που απαλλάχθηκαν από όλες τις κατηγορίες. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξή. Η διαδικασία τη συμφιλίωση και τη ομαλοποίηση των σχέσεων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων είναι θεμελιώδης συνθήκη για να υπάρξει μια επιτυχής πορεία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των συμφέρων της Σερβίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να συνεχιστεί η διαδικασία αυτή παρά τις αποφάσεις του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου. Το γεγονό είναι πως συνέβησαν εγκλήματα πολέμου στη Σερβία και Κουσφοπέδιο και πρέπει να καταδικαστούν από τα εγχώρια δικαστήρια στις χώρες αυτές οι δράστες. Επιπλέον υπάρχουν πάνω από 10.000 αγνοούμενοι από τα δεκαετία του 1990. Το ζήτημα αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει άπαξ και Η Σερβία έχει φτάσει το σκοντά όσο ποτέ στις ε, διαδικασίες έναρξης ε, των διαπραγματεύσεων ένταξη και ενθαρρύνουμε με τη σημερινή έκθεση την Σερβία και τους πολίτες της. Ελπίζω το Συμβούλιο σύντομα να είναι σε θέση να δώσει Σερβία μια ημερομηνία για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε την ε, Σερβία και βεβαίως θέλω να ευχαριστήσω και την γραμματεία της Επιτροπής μας και τους βοηθούς μας. Και αναμένω βεβαίως τις συζητήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κατσίν. Τώρα θα ήθελα να προτείνω το εξή. Επειδή ο χρόνος πιέζει και επειδή σχετίζεται και η επόμενη έκθεση με αυτό το θέμα, του κοσμοπεδίου δηλαδή, αν συμφωνούν οι δύο εισηγητές να τα δούμε μαζί. Αντιλαμβάνομαι πως ε, κυρία Λοχμπίλη αντικαθιστά την κυρία Λούνατσεκ. Σας δίνω λοιπόν το λόγο για να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις για το κοσμοπέδιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Λούνα Τσεκ μου ζήτησε να την εκπροσωπήσω γιατί να εκπροσωπήσω γιατί είναι άρρωστη. Θα ήθελα λοιπόν να παρουσιάσω κάποια σημεία της έκθεσης πρώτα απ' όλα. Η κυρία Λούνα Τσεκ ζήτησε να πούμε πως οπωσδήποτε υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα τα οποία θα ήθελε να πει, αλλά πρέπει να τηρήσει τους κανόνες. Οπότε οι εξηγήσει δεν είναι επαρκείς και ελπίζει να υπάρξουν αρκετές τροπολογίες για να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν η έκθεση καλωσορίζει το αποτέλεσμα της μελέτης σκοπιμότητας της Κομισιόν που είναι πως μπορεί να υπάρξει μία συμφωνία σύνδεσης με το κοσμοπέδιο όταν ε, ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των κρατομονών όσον αφορά το καθεστώς του κοσφοπεδίου. Αυτό είναι θετικό. Επίσης η έκθεση λαμβάνει υπόψη το ότι 10 Σεπτεμβρίου 2010 τελείωσε mm. η ανεξαρτησία υποεπιτήρηση καθώς η Διεθνής Ομάδα διατύπωσε πως ε, ε, εφαρμόστηκαν όλες οι συστάσεις για τον καθορισμό του καθεστώτος της χώρας αυτής. Επίσης η έκθεση χαιρετίζει τον ε, διάλογο υψηλού επίπεδου μεταξύ Πριστίνας και Βελιγραδίου που έδωσε νέα ορμή στις σχέσεις και επίσης ξεκαθαρίζει η έκθεση πως δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν παράλληλες δομές ή να συνεχίσουν να εφίσετε. Κατόπιν. η έκθεση χαιρετίζει ρητός την ε, εξέταση και την συνέχιση της εντολής της EULEX. Επίσης, ε, η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για την στήριξη για το κράτος δικαίου στο Κοσφοπέδιο, θέτει σημαντικά ερωτήματα και ζητάει από όλους τους ενδιαφερόμενους να εφαρμόσουν αυτά τα οποία αναφέρει η έκθεση για να βελτιωθεί η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, υπάρχει ανησυχία καθώς ε, δεν υπάρχει επιτυχία στην καταπολέμηση της διαφοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και ζητάει από τις αρχές του Κοσφοπεδίου να ενισχύσουν την πολιτική βούληση για την καταπολέμηση της διαφοράς σε κορυφαίο επίπεδο. βεβαίω. αυτό δεν ισχύει μόνο για το Κοσμοπέδιο αλλά και για άλλε χώρες στην περιοχή των Βαλκανίων. Κλείνοντα στο σημείο 12 γίνεται λόγο για την κατάσταση των μειονοτήτων, εθνικών, αλλά και σεξουαλικών. Πρέπει να ληφθεί υπόψη όπως ήδη την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε στην Επιτροπή Ανθρωπινών Δικαιωμάτων μία συζήτηση για την κατάσταση των μειονοτήτων, ειδικά των Ρωμά. Και αυτό νομίζω πρέπει να μπει στην έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Λόχπιλερ. Τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον σκιοδησηγητή του ΕΛΚ για τη Σερβία, τον κύριο Σέρφλιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο ε, Κάτσιν, ο οποίος έχει κάνει θαύματα. Θα δείτε βεβαίως και τις τροπολογίες οι οποίες έχουν διανομηθεί. Θα ήθελα να δούμε θέματα αρχής καταρχήν ως προς τη Σερβία και το Κωσυφοπέδιο. Ε, η πολιτική και ο νόμος ε, κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Και αν δείτε το Σύνταγμα της Σερβίας βλέπετε ότι αναφέρει ότι το ε, Πέδιο είναι αναπόσπαστο τμήμα της Εθνικής Επικράτειας της Σερβίας. Αυτός ο νόμος που ισχύει στη Σερβία ε, αντιβαίνει αντιβαίνει τις πολιτικές κατευθύνσεις που επιθυμούμε εμείς για τη Σερβία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε. Θα πρέπει να εξωθήσουμε τη Σερβία σε συνταγματική αναθεώρηση. Είναι, ξέρω ότι είναι παράτολμο αυτό που λέω, αλλά κάποιος πρέπει να το πει. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ως προς την αυτονομία της Βοηβοδίνας, ε, αυτό αντιβαίνει μία προηγούμενη έκθεσή μας σε σχέση με την αποκέντρωση που είχαμε προτείνει στη Σερβία. Ως προς το κοσυφοπέδιο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι Σέρβοι του Κωσυφοπεδίου δεν ήθελαν την ηθαγένεια του Κωσυφοπεδίου. Δηλαδή, ό,τι και να συμβεί, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Άρα ας αναγνωρίσουμε την κατάσταση και ας τη ρυθμίσουμε. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Κάτι άλλο γενικότερο που ανακύπτει και από την έκθεση Κατσίν είναι η οικονομία. Η οικονομία Τη Σερβία είναι αξιολύπητη. 30% ανεργία, γενικά Σερβία 50% δείκτης ανεργίας για τους νέους. Ένα προς ένα σχέση εργαζομένων μη εργαζομένων. Μην ξεχνάμε βεβαίως και τα μεταναστευτικά ρεύματα και τις πιέσεις προς τις ευρωπαϊκές χώρες και κάτι άλλο. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει θα πρέπει να ζητήσουμε να ανοίξουν τα αρχεία ούτμπα της Σερβίας, διότι δεν είναι ένα θέμα της Σερβίας που αφορά τη Σερβία με το παρελθόν της, αλλά και όλες τις άλλες πρώην ομοσπονδίες της ε, Ιουγκοσλαβίας. Δηλαδή, οι εμπλεκόμενοι ε, φορείς θα πρέπει να ανοίξουν τα αρχεία, τα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών από το 45 και μετά. Ευχαριστούμε κύριε Σούπλιν, ιδιαίτερα για το τελευταίο θέμα που θίξατε, σύμφωνα απόλυτα. Η κυρία Κοπά, σκιώδης για τη Σερβία από πλευράς ε, σοσιαλιστών, για δύο λεπτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, δύο εισηγητές για τις εκθέσεις τους και συμφωνώ με τον κύριο Κάτσιν ότι είναι θετική έκθεση και αντικατοπτρίζει τη θέση ως προς τη Σερβία. Δηλαδή θα πρέπει να της δώσουμε ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων ως προς τις ε, τριπλές ε, εκλογές του παρελθόντος Μαΐου ήταν ύψης της σημασίας και καταλαβαίνω την παράγραφο 1 του εισηγητή όπου μιλάει για την σωστή διενέργεια των εκλογών. Είναι πολύ σημαντικό διότι γίνεται λόγος και για τις θετικές εξελίξεις. Όμως αυτό δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η επιτελέστηκε μικρή πρόοδος από το Μάρτιο 2012 όταν η Σερβία έλαβε το καθεστώς της υποψηφιότητας, θεωρήθηκε υποψήφια χώρα. Όπως είπε η κυρία Λούνατσεκ, η νέα κυβέρνηση μας είπε ότι θα συνεχίσει την διαδικασία ολοκλήρωσης, όμως αναμένουμε απτά αποτελέσματα. Καλό το μήνυμα, αλλά έμπρακτα τι γίνεται. Χρειαζόμαστε κάτι έμπρακτο, ιδιαίτερα μετά στις 100 μέρες της διακυβέρνησης. Είναι γεγονός ότι γίναν πολλές διαπραγματεύσεις ε, για να δημιουργηθεί η κυβέρνηση και βεβαίως και με το καλοκαίρι ε, επιβραδύνθηκε η διαδικασία και δεν θα μπορέσει μάλλον να αποφασίσει το Συμβούλιο ότι το Δεκέμβριο για την έναρξη διαπραγματεύσεων ακόμα και εάν στο μεταξύ εξομαλυνθούν οι σχέσεις με την Πρίστινα. Αυτό το λέω γιατί όταν συζητούσαμε στο Βελιγράδι με την κοινωνία των πολιτών, κατά τις συζητήσεις αυτές αναφέρθηκε το γεγονό ότι τονίζουμε υπερβολικά το κοσυφοπαίδιο και δεν ασχολούμαστε επαρκώς με την, τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Θα πρέπει να ακούσουμε αυτό, το, αυτή την αιτίαση και γι' αυτό το σχέδιο έκθεσης αφιέρωσε μία έκθεση Αλλά τώρα βλέπω ότι υπάρχει μια ολόκληρη σελίδα για το κοσυφοπαίδιο και δεν χρειάζεται να επαναλαμβανόμαστε. Δεν νομίζω θα υπάρξουν ε, μείζονες αποκλήσεις ως προς τις προοπτικές. Θα ήθελα αυτή η έκθεση να παραμείνει μια έκθεση που να αφορά τη Σερβία και όχι να εμπλέκεται το κοσυφοπέδιο. Δηλαδή να έχουμε μια μικρότερη παράγραφο επί του θέματος. δεν είναι έκθεση που αφορά το κοσυφοπέδιο, διότι αυτό θα ήταν ένα λανθασμένο ε, μήνυμα προς τους Σέρβους. Χρειάζονται, χρειάζεται εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτερα, ιδιαίτερα το δικαιοδοτικό προς το δικαιοδοτικό, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τις διάφορες ελευθερίες. η διαχωριστική γραμμή μεταξύ πραγματικής καταπολέμησης ε, είναι, δεν είναι τόσο ε, εύκολα ορατή, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για απομάκρυνση πολιτικών αντιπάλων μέσα στα πλαίσια της δίθεν καταπολέμησης της διαφθοράς. Δεν θα προχωρήσω περαιτέρω. Θα σταματήσω, θα σταματήσω. Θα έχουμε άλλη ευκαιρία συζήτησης. Ευχαριστώ το Γέλκο Κάτσι και την ε, κυρία Λούνετσεκ ε, γιατί αποστέλουν θετικά μηνύματα για τη διαδικασία διεύρυνση στην ε, περιοχή. Ούτε 15 λεπτά δεν έχουμε συνάδελφοι και πολλοί θέλουν το λόγο. Ο κύριος Τάνοκ που είναι σκιώδης για τις εκθέσεις Σερβίας Κωσυφοπεδίου. Αυτά είναι οι αρετές της μικρής ομάδας. Αλλά είμαι και εισηγητής για το Μαυροβούνιο. Ευχα... Συγχαίρω λοιπόν... Α, πώς τι... Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κάτσιν για την παράγραφο 22 που μιλάει για βελτιώσει σχέσεων Σερβίας και Μαυροβουνίου. Την παράγραφο 5 για τη συνεργασία της Σερβίας με το Διεθνές Δικαστήριο και τον διάλογο Πριστίνης και Βελιγραδίου. Επίσης ημερίζομαι την καταδίκη της απαγόρευσης του Gay Parade. Γιατί προφανώς δεν συμφωνεί, δεν συμβαδίζει με τη μοντέρνα σκέψη. Ελπίζω να ακυρωθεί. Εξάλλου δεν συμφωνεί και με αυτά που απεφάσισε το γειτονικό Μαυροβούνιο. Το άρθρο 359 μιλά για ορισμένες διακοσμητικές μονοαλλαγές. Εγώ έχω αγγλοσέρβους ψηφοφόρους που θεωρούν ότι χρησιμοποιείται η διάταξη αυτή για να τους ζημιώσει. Είναι φαίνεται κατάλοιπα του κομμουνιστικού παρελθόντος. Γι' αυτό καταδικάζω τη χρήση του 359 από τη σερβική κυβέρνηση που δεν έχει θέση σε μια μοντέρνα χώρα. Κατά τα άλλα χαίρομαι ιδιαίτερα για την έκθεση αυτή και συγχαίρω τη Σερβία για την υποψηφιότητά σας για την έκθεση Λούνατσεκ. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι δουλειά του Κοινοβουλίου μας να κρίνει αυτά τα πράγματα για την αναγνώριση μη του κοτσιφοπεδίου δηλαδή. Είναι δικό τους θέμα. Το θέμα της αναγνώρισης του ημί είναι πολύπλοκο νομικό θέμα, καθώς και ο χωρισμός του κοσυφοπεδίου είναι θέμα που παραμένει ανοιχτό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ. Τώρα ο κύριος Κούκαν που είναι πρόεδρος της Επιτροπής για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Είναι κρίμα το ότι έχουμε τόσο λίγο χρόνο. Για την έκθεση για τη Σερβία θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το σχέδιο Κάτσιν. Θεωρώ πως είναι αντικειμενική, θετική έκθεση η οποία εκτιμά θετικά τη διαδικασία ολοκλήρωσης με τη Σερβία και στέλνει τα σωστά μηνύματα. Επίσης στηρίζω πλήρως την έκκληση προς την Κομισιόν για να δοθεί ημερομηνία για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Βεβαίω δεν θα γίνει αυτομάτως. Η Σερβία θα πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις ε, και όλα τα σχετικά. Θεωρώ πως είναι σημαντικό να αναφέρουμε την καταπολέμηση της διαφθοράς οργανωμένου κλίματος, στο άρθρο 359, ε, διάσημο ή διαβόητο. Τα έχει αναφέρει αυτά ο κύριος Κατσίν. Ε, πράγματι, θεωρώ πως θα παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις για την περιφερειακή συνεργασία, νομίζω η Σερβία τα πάει καλά. Αξίζει νομίζω να υποθούν λίγο περισσότερα λόγια. Επίσης πρέπει να δοθεί έμφαση στη διαδικασία συμφιλίωσης, ειδικά μετά τα όσα, τις τρεις τελευταίες αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Εγώ θεωρώ πως αυτά είναι τεστ για το σερβικό λαό και τη σερβική ηγεσία κρίνοντας από τις δηλώσεις ε, και συμπεριφορά των κορυφαίων Σέρβων ηγετών συμπεριφέρονται με τρόπο υπεύθυνο και φιλοευρωπαϊκό και αυτό είναι κάτι το ενθαρρυντικό. Θεωρώ λοιπόν πως αναμένουμε εδώ συνεργασία με τον κύριο Κατσίν για την, τελική μορφή του ψηφίσματος. Ήταν πάρα πολύ καλή δουλειά που έγινε και δεν τα λέω αυτά τυπικά για το κοσφοπέδιο. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Λούνατσεκ για την καλή τη έκθεση. Δεν τίθεται ζήτημα πω το κοσφοπέδιο έχει επιτύχει πρόοδο. Η μελέτη σκοπιμότητα τη Κοντουσιών ανοίγει την πόρτα για περαιτέρω βήματα με το κοσφοπέδιο. Καλωσορίζω αυτό το οποίο λέει η Κομισιόν, που στα τελευταία τρία χρόνια το Κοσμοπέδιο έχει αυξήσει τη δυνατότητα εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ε, συμφωνίες. Μην χτυπήσετε το σφυράκι σας παρακαλώ. Το σχέδιο έκθεσης ε, αναφέρει σαφώς αυτά τα ζητήματα, ειδικά αυτά τα οποία πρέπει να ε, οριστικοποιηθούν ακόμα, αναφέρεται η απελευθέρωση και τα λοιπά, να σταματήσει δηλαδή η απομόνωση του κοσφοπεδίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει πολλά στο κοσφοπέδιο και η διαδικασία ένταξης θα πρέπει να συνεχίσει. Είναι σημαντικό ε, το ότι το ελεγκτικό συνέδριο έκανε μια έκθεση. Δεν συμφωνώ με αυτό το οποίο επισημαίνεται. Ε, δηλαδή συγκεκριμένε δυσκολίε λόγω της μη αναγνώρισης 5% μελών. Συμφωνώ πως αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, αλλά δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Επίσης θεωρώ πω κάποιες παράγραφοι θα χρειαστούν μεγαλύτερη ε, προσοχή για να έχουμε πιο ισορροπημένη διατύπωση, ειδικά αυτές που αφορούν τις σχέσεις ε, Σερβίας-Κοσφοπεδίου. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε κύριε Κόκαν και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Πόσελ ο οποίο είναι σκιώδης ηγητής για την ομάδα του ΕΛΚ για το Κοσφοπεδίο. Ναι κύριε Πρόεδρε, θέλω να στηρίξω αυτά τα οποία είπε η κυρία Λούνατσεκ πρέπει να ενισχυθούν και όλα. Σημαντικότερα εδώ πέρα είναι βεβαίως ε, το ότι αρνούμαστε οποιαδήποτε διαμπελισμό του κοσμοπεδίου, καθώς να δεν μπορεί να οδηγηθούμε πάλι σε ενοπλές συγκρούσεις. Και θα πρέπει επίσης η Σερβία να δούμε και το θέμα της κοιλάδας του Πρεσέφου. Μετά θα μπουν και άλλες χώρες ε, στη Διαμάχη, Μαυροβούνιο, Πουγκουδουμού και θα ανοίξουμε τον ασκό του αιώλου. Τα έχουμε πει πολλές φορές, επικυρώσει με πλειοψηφία τριών τετάρτων, εδαφική ακεραιότητα του κοσφοπεδίου με προστασία των μειονοτήτων. Και αυτό αναφέρεται και στο Σύνταγμα των Κωσοβάρων και το σχέδιο Αχτισάρη νομίζω πως είναι το καλύτερο στα Δυτικά Βαλκάνια αλλά ε, βεβαίως δεν γίνονται αρκετά πράγματα στην πράξη αλλά θεωρητικά ε, είναι μια χαρά. Ε, υπενθυμίζω το πέρα το Πρέσεβο ως παράδειγμα για τους Σέρβους. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ε, τα ίδια μέτρα και στάθμα για τις δύο χώρες. Καλύτερο θα ήταν βεβαίως μια διμερή συμφωνία στην οποία και οι δύο χώρες θα εφάρμοζαν τα ίδια πράγματα για τις μειονότητες τους. Αλλά από κάτι τέτοιο απέχουμε ακόμα πολύ. Γι' αυτό θεωρώ πως οι διατυπώσεις στην έκθεση Κατσίν για τις μειονότητες ε, είναι θετικές. Πρέπει να προσπαθήσουμε να μετράμε τις δύο χώρες με τα ίδια μέτρα. Μόνο έτσι θα μας πάρουν και σοβαρά γι' αυτό, λέω ξεκάθαρα, στήριξη για αυτά τα οποία λέει η κυρία Λούνατσεκ, στήριξη και για την έκθεση του κύριου Κατσίν, όσον αφορά όμως συνταξιακές διαπραγματεύσεις και τις μειονότητες, εγώ είμαι υπέρ του να κάνουμε λίγο πιο ήπια τη διατύπωση. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε κύριε Πόσελτ. Θα δώσω λόγο στον κύριο Παντσέρη που είναι ισχυρός ζητή. Ε, εντάχει, η έκθεση αυτή είναι μεταβατική και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, γιατί πρόκειται για μία μακροχρόνια διαδικασία. Έχουμε να κάνουμε με μία πραγματικότητα που αφορά καταρχήν την ανεξαρτησία και την εθνική κυριαρχία, την ενίσχυση της κυριαρχίας με μεταρρυθμίσεις ολοένα και μεγαλύτερες και υπάρχει μια διαφορετική πραγματικότητα που αφορά το ρόλο της ε, διεθνούς κοινότητας και ένα τρίτο πιο προβληματικό επίπεδο που αφορά την κοινότητα αυτή του Βορείου Κωσυφοπεδίου. Νομίζω ότι η έκθεση θα πρέπει να είναι πιο στεναρή δηλαδή μεταρρυθμίσεις και διάλογος θα πρέπει να είναι πιο άρρηκτα συνδεδεμένοι. Και τους προσεχείς μήνες είτε η διεθνής κοινότητα είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ορίσουν μεγαλύτερη σαφήνεια σε αυτά τα τρία επίπεδα. Και ζητηθεί ε, προσέγγιση όχι μόνο από πλευράς ε, Σερβίας, αλλά και από πλευράς ε, Κωσυφοπεδίου, να ζητηθεί μια σύγκληση στην προσέγγιση αυτή. Τέσσερις ομιλητές ζήτησαν το λόγο. Ένα λεπτό καθένας. Αυτή η συζήτηση για επόμενη για την Ισλανδία θα πρέπει να ε, αναβληθούν. Έπεσαν θύμα στο βωμό της Αιγύπτου, Λανσβέργης. Δεν ζητήσατε το λόγο κύριε Λανσβέργης. Ο κύριος Πρέντα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Και εγώ ήθελα να ζητήσω να θα αναβληθεί η συζήτηση για την Ισλανδία και να λάβουμε υπόψη ότι θα ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις με τη Σερβία το συντομότερο δυνατόν. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν ορισμένες αντιφατικές έννοιες γιατί να δεν ζητήσαμε την αναγνώριση της ανεξαρτησίας, αλλά έμπρακτα θέλετε να συμπεριφερθεί η Σερβία σαν είχε ήδη προβεί στην αναγνώριση. Δηλαδή να μην υπάρχουν παράλληλες ε, υποδομές του Βορείου Κωσυφοπεδίου. Ζητάμε να αποσυρθούν από το Βελιγράδι. Δηλαδή πώς θα γίνει αυτή η ομαλοποίηση των σχέσεων με το κοσυφοπέδιο πριν από την απαρχή των ε, διαπραγματεύσεων. Τι θα πει στην ουσία αυτή η διαδικασία, τι σημαίνει έμπρακτα αυτή η διαδικασία για αυτή την υποψήφια χώρα. Uh, Ευχαριστούμε κύριε Πρέδα, ο κύριος Κυρία, ευχαριστώ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και γι' αυτό πρέπει να είμαι σύντομη γιατί δεν θέλω να επαναλάβω. Νομίζω ότι στο κείμενο ε, του κύριου Κάτσιν και της κυρίας Λούνετ ε, και τα λέει όλα. Όλα. Όλα. Ο κύριος Κούκαν, επαναλαμβάνω, τα είπε όλα και συγχαίρω τον Γέλκο που μπόρεσε να συμπεριλάβει όλα αυτά τα στοιχεία στην έκθεση του εξαιρετικό, εξαιρετικό. Επίσης συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν για τις τρεις καινούργιες παραγράφους και ίσως και εγώ να καταθέσω μερικές τροπολογιούλες αλλά γενικά, γενικά λέγω, εξαιρετική η έκθεση. Ελπίζω μόνο η κυβέρνηση να εφαρμόσει όλα όσα ζητάμε. Τελευταίος ο κύριος Πέτερλε. Ευχαριστώ. Η κατάσταση στην περιοχή είναι πολύ δύσκολη, τεταμένη και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε μια εξέλιξη, κάποιες εξελίξεις εκεί εξελίξεις. Υπήρξε πρόοδος βέβαια στη Σερβία, αλλά χαίρο τον εισηγητή γιατί χρησιμοποίησε το σωστό ύφος. Λοιπόν, τον σωστό τόνο. Χαίρομαι επίσης που η Σερβία προσεγγίζει το κράτος δικαίου και έχει περισσότερο διάλογο με την Πρίστινα. Σε άλλα θέματα βέβαια δεν διαπιστώνεται πρόοδος γιατί συνεχίζουν να υπάρχουν εσωτερικές διαφωνίες. Διακρίνει κανείς κάποια πιο φιλοευρωπαϊκή στάση στη Σερβία αλλά νομίζω ότι οι πολιτικοί, οι Σέρβοι πολιτικοί θα ακούσουν επιτέλους το μήνυμα των Βρυξελών. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πέτερλε και τώρα μήπως η Κομισιόν για την πιθανή διεύρυνση, Είναι πολύ σύντομα ήθελα να ευχαριστήσω τους συζητητές συμφωνούμε και εμείς η Σερβία πρέπει να εφαρμόσει αυτά που υποσχέθηκε και τις καλές της προθέσεις. Αρχίζει επιτέλους να το πράττει, οι μεταρρυθμίσεις αρχίζουν σε πιο σταθερό ρυθμό και θα υπάρξει σε λίγο ένα σχέδιο δράσης και εθνικό σχέδιο για την εφαρμογή του κεκτημένου. Όλα αυτά μπορεί επίσης να τα πείτε στην έκθεσή σας γιατί είναι βήματα που θα υλοποιηθούν σε λίγο. Και πράγματι βασίζονται στην υλοποίηση των υπολείπων μετά. Η Σερβία ελπίζει να αρχίσουν σύντομα οι διαπραγματεύσεις εφόσον βέβαια βελτιωθούν ουσιαστικά οι σχέσεις με το κοτσιφροπέδιο. Πρέπει να διαχωρίσουμε σαφώς τι χρειάζεται να γίνει σε αυτήν τη φάση. Και είναι οι κύριες προτεραιότητες που καθορίστηκαν πέρυσι. Και κάναμε και ένα διαχωρισμό με το, την πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση που χρειάζεται για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το κοτσιφοπέδιο. Γι' αυτό Απαιτείται μία βήμα-βήμα προσέγγιση και γι' αυτό το περιλάβαμε μεν στις διαπραγματεύσεις αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα υπάρξει ουσιαστική πρόοδο στην επόμενη περίοδο. Το σημαντικό τώρα θα ήταν ο υψηλού επίπεδου διάλογος να φέρει νέα αποτελέσματα ιδιαίτερα την εφαρμογή των συμπεφωνημένων και θα το παρακολουθούμε από κοντά. Θα γράψουμε έκθεση όταν θα υπάρξει ουσιαστική πρόοδος. Η δική σας έκθεση του Μαρτίου θα είναι πολύ επίκαιρη. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Τώρα για το κοτσιφοπέδιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λούνατσεκ. Και να ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση. Δύο πράγματα μας απασχολούν. Όπως ε, αναφέρθηκε στη μελέτη αντικτύπου, θα θέλαμε να υπάρχει ένα προσχέδιο διαπραγματεύσεων με το Κωσυφοπέδιο με βάση τις προτεραιότητες που ορίσαμε για το Κωσυφοπέδιο και παράλληλα την ε, συνέχιση του πολιτικού διαλόγου υψηλού επίπεδου διότι θα έχει μεγάλες επιπτώσεις στις σχέσεις και στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κωσυφοπεδίου και ελπίζουμε αυτό να αντικατοπτρίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Κάτσιν και Λόχμπίλερ. Εντάχει γιατί πρέπει να κλείνουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα θετικά που ακούσαμε μεταξύ μας εδώ πέρα. Πρέπει και τη Σερβία και το Κοτσιφοπέδιο να τα αντιμετωπίσουμε θετικά, με θετικό πνεύμα. Ήθελα απλώς να μιλήσω για μερικά πράγματα που υπόθηκαν εδώ. Πρώτον, σας πληροφορώ ότι όλοι οι σκιώδεις έχουν πολύ μακρύτερες εκθέσεις και πληρέστερες και η κατάθεση τροπολογιών θα συνεχίσει. Όσο για αυτά που είπε ο κύριος Πόσελτ για τα θέματα μειονότητων στη Σερβία, νομίζω ότι και αυτά ήταν σωστά. Δεν είναι δικιά μου δουλειά βέβαια αυτό. Εγώ υπέβαλα το σχέδιο αλλά ελπίζω και εσείς να καταθέσετε. Άλλο τώρα. Αυτά που ζήτησε η κυρία Κόπα αλλά που είναι από τη χώρα που δεν αναγνωρίζει το Κότσοβο. Εδώ μας μίλησε για ευσεβείς πόθους. Στη Σερβία δίνουν πολύ μεγαλύτερο χώρο για τις ειδήσει από το Κωσυφοπέδιο από ό,τι μαζί ζήτησε εκείνη. Τι είναι εδώ πέρα, παράπλευρες απώλειες. Από την άλλη, αυτό που εξέπληξε τη Σερβία και είναι εδώ το σχόλιο μου προς τον κύριο Τάνοκ που αναμένει πέντε ακόμη χώρες να αναγνωρίσουν το κοσυφοπαίδιο. Αυτές οι πέντε χώρες αντιτίθενται και στη διαμέληση του κοσυφοπαιδίου. Η Σερβία κατανοεί αυτό το πράγμα και έτσι διευκολύνονται τα πράγματα. Αύριο θα συναντήσω τον κύριο Θάτσι και τον κύριο Ντάτσιτς γιατί είμαστε σε συνεχή διάλογο μαζί τους και πιστεύω ότι με την ενεργή τους συμμετοχή σε αυτόν τον διάλογο κάνουμε πραγματική πρόοδο. Εδώ δημιουργούμε την αμοιβαία εμπισουτοσύνη και δεν πρέπει να συζητάμε μόνο την αξιολόγηση ως προς την κυβέρνηση. Υπάρχουν δύο προβλήματα. Ο πρόεδρος της Σερβίας δεν πήγε να δει όλους τους γείτονές του και ελπίζω να ταξιδέψει πιο πολύ, ιδίως στην Κροατία. Και το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετάσχει στον διάλογο εκεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. κατάλαβα ότι η έκθεση Λούνα Τσεκ την χάνει ευρεία εμπιστοσύνη και θα διαβιβάσω τα σχόλια απευθείας σε εκείνη. Έχουμε και δύο εκθέσεις πολύ σημαντικές, θα τις αναβάλουμε. Προθεσμία τροπολογιών 9 Ιανουαρίου για τη Σερβία και για το Κωσυφοπέδιο και για τις δύο εκθέσεις. Αναβάλλεται το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης για μια προσεχή συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Χαίρετε.